<clears throat> Euh, Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Η σημερινή μας συνεδρίαση πρωινή θα αφιερωθεί κυρίως στο θέμα του διαστήματος. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς την ημερήσια διάταξη. Καταρχάς, για μία ώρα περίπου, μία ώρα και ένα τέταρτο το πολύ, θα ασχοληθούμε με την διαστημική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά υπό το πρίσμα της ασφάλειας και άμυνας. Γιατί για πρώτη φορά, όπως ξέρετε, με τη συνθήκη της Λισαβόνας γίνεται ρητή μνήα μιας ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής. Σε ένα από τα άρθρα, το διατακτικό της συνθήκης της Λισαβόνας. Οπότε ήδη έχουν ξεκινήσει διάφορες συνεργασίες και μπορούν περαιτέρω να εξελιχθούν. Οπότε το θέμα τα ασφάλειας και άμυνας στα πλαίσια της διαστημικής πολιτικής είναι πολύ σημαντικά. Γιατί θα εξασφαλίσουν μια πραγματική στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως ε, Ο λόγος της α, ε, μικρής προσέλευσης σήμερα οφείλεται στη σύμπτωση της σημερινής μας συνεδρίασης με μια συνδιάσκεψη για το διάστημα που το διοργανώνει Business Bridge Europe υπό την αιγίδα του Πρόεδρου Μπούζεκ. Είναι μια διήμερη συνδιάσκεψη για το διάστημα και η αυριανή μάλιστα ημέρα θα αφιερωθεί σε θέματα διαστημικής πολιτικής ε, για υπό το πρίσμα πάλι της ασφάλειας και της άμυνας. Ίσως γι' αυτό έτσι εξηγείται η μικρή παρουσία. Έχουμε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την κυρία Κάνης Χιούμπερ από την μονάδα της Ιδιαστημικής πολιτικής και του συντονισμού. Έχουμε την κυρία Νάζα από, την, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, επιφορτισμένη με τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κύριο Πάρης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, υπεύθυνο για, το για το σχέδιο SATCOM και το Space Situational Awareness για την επαγρύπνηση ως προς την θέση στο διάστημα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ε, θα ακούσουμε πρώτα τις δικές σας εισηγήσεις και μετά θα γίνει μια μικρή συζήτηση με τους παρόντες. Θα ακούσουμε πρώτα την κυρία Χατσμέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Ντονζόν και καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι αρκετά νωρίς το πρωί. Λέγομαι Σίλβια Κάινς Χούμπερ και είμαι τμήματάρχης της ε, Μονάδας Διαστημικής Πολιτικής και Συντονισμού των ε, Δραστηριοτήτων Διαστήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση σήμερα το πρωί, χωρίς διεξοδική ανάλυση γιατί είχαμε πολλές ε, παρουσιάσεις και δώσαμε πολλές εξηγήσει για την Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική. Εγώ θα επικεντρωθώ στις αλλαγές και στις επιπτώσεις ε, που έχει η συνθήκη της Λισαβόνας, η νέα συνθήκη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο συγκεκριμένα 189 που αφορά τις ε, αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το διάστημα. Θα δούμε λοιπόν τις επιπτώσεις της συνθήκη στη διαστημική πολιτική, θα δούμε τις αλλαγές στην κατάσταση και θα επισέλθω σε κάποιες λεπτομέρειες στα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Υπό το πλαίσιο φυσικά του νέου νομικού πλαισίου, υπό πρίσμα του νέου νομικού πλαισίου και του άρθρου 189. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας η διαστημική πολιτική έγινε μια αυθυπόστατη πια ευρωπαϊκή πολιτική. Πρόκειται για κοινή αρμοδιότητα ή παράλληλη αρμοδιότητα, κάτι που σημαίνει ότι η κοινοτική αρμοδιότητα, η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα δεν ε, εμποδίζει τα κράτη-μέλη να ασκήσουν τις δικές τους αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, η ευρωπαικη αρμοδιοτητα δεν εμποδιζει τα κρατη μελη να ασκησουν τι δικε του αρμοδιοτητε σε εθνικο επιπεδο ταυτοχρονα η συνθηκη τη Λισαβόνα δίνει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολιτική ταυτότητα για θέματα διαστήματο και με βάση την ερμηνεία μα για το άρθρο 189 συνδέει η συνθήκη το διάστημα με την εφαρμογή πολλών κοινοτικών πολιτικών. Έτσι το διάστημα η διαστημική πολιτική συνδυάζεται με την εφαρμογή πολιτικών που σχετίζονται με τη νέα ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ήδη με κάποιους τρόπους πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει τις ε, νέες ή τις ενισχυμένες αρμοδιότητες για θέματα πολιτικής διαστήματος σε ό,τι αφορά τη χάραξη μια νέα διαστημική πολιτική, η συνθήκη αναφέρεται σε κοινέ πρωτοβουλίε ε, για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και στη δυνατότητα συντονισμού των προσπαθειών που χρειάζονται για την εξερεύνηση και την ε, εκμετάλλευση του διαστήματος. Το άρθρο 2.4 προβλέπει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Οπότε αν συνδυάσουμε τα δύο άρθρα 2.4 και 189 μπορούμε να ερμηνεύσουμε το άρθρο 189 ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δραστηριότητες μας στο διάστημα για την εξυπηρέτηση της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Βέβαια αυτή είναι η δική μας ερμηνεία με τη βοήθεια φυσικά της νομικής υπηρεσίας, γιατί εγώ προσωπικά δεν είμαι νομομαθής. Επανέρχομαι λοιπόν στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας που προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θεσπίσει κάποια μέτρα για να εφαρμόσει τις αρμοδιότητές της και κάτι τέτοιο μπορεί να λάβει τη μορφή ακόμη και ενός ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος. Κάτι άλλο που προβλέπει η συνθήκη είναι ότι ήδη υπάρχουν προκαθορισμένε σχέσει με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματο, αλλά αυτέ τι ε, ήδη υπάρχουσες σχέσει τι θεσμοποιεί, ουσιαστικά τι επισημοποιεί η συνθήκη τη Λισαβόνα, θεσπίζοντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταρτήσει τις ε, κατάλληλες σχέσεις με, την με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Δεν αρχίζουμε δηλαδή εκ του μηδενός. Η ΕΣΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια, έχει πολύ σημαντικές αρμοδιότητες σε θέματα διαστήματος, ε, ερευνητικών προγραμμάτων, προγραμμάτων τεχνολογικής ανάπτυξης και εφαρμογή προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται σε μεταγενέστερο στάδιο και σε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, εθνικές πολιτικές. Έχουμε και μια συμφωνία πλαίσιο με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος από το 2004 που ήδη μια φορά ανανεώθηκε, παρατάθηκε και αυτή τη στιγμή ισχύει μέχρι το 2012. Οπότε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο ΕΣΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, είναι πολύ χρήσιμος, ανεκτήμητος. Και από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας με τη Συμφωνία Πλαίσιο είχαμε πολύ θετικές εμπειρίες από τη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Τώρα θα δούμε πώς θα ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία με τις νέες μας αρμοδιότητες από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Πάντως, ως σημείο αφετηρίας, αποστολή μας ε, θα ήταν η ενίσχυση αυτών των σχέσεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, συνεχίζοντας ε, το πολύ αξιόλογο έργο της του ΕΣΑ εδώ και 40 χρόνια σε συνδυασμό με τις νέες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προκύπτουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ας δούμε τώρα τα πρώτα βήματα μετά από την εισαγωγή της συνθήκης. Ήδη έχουν γίνει κάποια πρώτα βήματα σε επίπεδο διακυβέρνησης ό,τι αφορά τη διαστημική πολιτική στο στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει προβλέψει και ένα σχηματισμό συμβουλίου για το διάστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποφασίστηκε η συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας για τις νέες διαστημικές δραστηριότητες. Μάλιστα αυτή τη στιγμή συγκροτείται η ομάδα εργασίας και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεδριάσει για πρώτη φορά τις επόμενες εβδομάδες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή αναλύει και τη δική της στρατηγική, την πρόταση που θα υποβάλει για το τι μορφή θα λάβει η διαστημική ευρωπαϊκή πολιτική στο μέλλον. Βέβαια δεν ξεκινούμε εκ του μηδενός. Ήδη οι προεδρίες, οι προηγούμενες έχουν θέσει κάποιες προτεραιότητες και οι Υπουργοί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε προηγούμενα ψηφίσματά του έχουν ε, δηλώσει τις προτεραιότητές τους για το διάστημα. Μυστικά δεν υπάρχουν. Καταρχήν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την συνέχιση των δύο σημαντικών προγραμμάτων στο μέλλον, του Γαλιλαίου και του GMS, του προγράμματος γεωσκόπησης. Και φυσικά, επειδή υπάρχουν πολύ σημαντικοί εταίροι στο διάστημα, θα πρέπει να θεωρήσουμε τις ε, υποδομές μας για τη διαστημική πολιτική ως κέρυες κρίσιμες υποδομές και να τις προστατεύσουμε φυσικά. Επίσης, το θέμα της ασφάλειας και του διαστήματος είναι μια τρίτη προτεραιότητα που θα πρέπει να τη συμπεριλάβουμε στη διαστημική πολιτική του μέλλοντος. Θα επανέλθω αργότερα στο θέμα αυτό, ποιες είναι οι προθέσεις μας δηλαδή και ποια η βασική μας κατεύθυνση. Και τα τελευταία χρόνια, στο θέμα της εξερεύνησης του διαστήματος, και η εξερεύνηση του διαστήματος είναι σημαντικό θέμα. Μόλις πρόσφατα έγινε μια συνδιάσκεψη γι' αυτό με θέμα τι μπορεί να προσφέρει εδώ εκτός από την τεχνογνωσία της Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχουμε φυσικά και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και πολιτικές αρμοδιότητες και μπορεί να αναβαθμίσει την εξερεύνηση του διαστήματος και να τις να προσδώσει και έναν πολιτικό χαρακτήρα. Ήδη εδώ και ένα χρόνο έχουμε σχετικές ε, συζητήσεις και ήδη σε μια συνδιάσκεψη που έγινε την τελευταία εβδομάδα με τους διεθνείς μας εταίρους καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα όπως ότι πρώτο βήμα είναι να δημιουργηθεί μια διεθνής πλατφόρμα υψηλού επίπεδου όπου θα συνεργαστούμε με τους ε, διεθνείς μας εταίρους για θέματα εξερεύνησης του διαστήματος. Τώρα, ως προς, τις, ε, ως προς την πορεία μας, τη μελλοντική μας πορεία για θέματα διαστήματος και άμυνας και ασφάλειας μάλλον. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνει πιο ισχυρός εταίρος σε θέματα διαστήματος, καταρχήν ήδη έχουμε το ίγνος, ε, πρωτοστατούμε στο πρόγραμμα Γαλιλαίος και θα έχουμε την ιδιοκτησία στα επιτεύγματα του Γαλιλαίου. Επίσης έχουμε και το πρόγραμμα GMES της ε, Ευρωπαϊκής Γεωσκόπησης. Θέλουμε να, να μεταθέσουμε αυτό το πρόγραμμα με τον πρόσφατο φαρμαστικό κανονισμό σε ένα επιχειρησιακό επίπεδο, σε μια επιχειρησιακή φάση. Επίσης, ό,τι αφορά το δορυφορικό πρόγραμμα, ε, βρίσκεται υπό επεξεργασία και βέβαια το θέμα είναι ποιος θα θεωρηθεί ο ιδιοκτήτης αυτών των constellation, των satellite constellation. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ο βασικός ιδιοκτήτης αυτών των ε, ε, ομάδων δορυφόρων και φυσικά θα φέρει την ευθύνη της προστασίας των υποδομών αυτών στο μέλλον. Φυσικά και οι Υπουργοί των Κρατών Μελών μα ζητούν να λάβουμε τα μέτρα και να θεσπίσουμε την σωστή προστασία για τις υποδομές αυτές. Μία συγκεκριμένη δραστηριότητα στον τομέα αυτό είναι να έχουμε μια ευρωπαϊκή πραγματικά δυνατότητα, ένα ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης των περιουσιακών μας στοιχείων για να ξέρουμε να πάση στιγμή ποιες είναι οι διαθεσιμάρχουν τέτοιες τέτοιε ικανότητες, τέτοιο δυναμικό σε εθνικό επίπεδο, αλλά φυσικά θα πρέπει τέτοιες υπηρεσίες να προσφέρονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί παραλαμβάνω θα δημιουργηθούν και ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία πέραν των εθνικών. Οπότε θα πρέπει να έχουμε και ένα ευρωπαϊκό σύστημα ετοιμότητες. Ο κύριος Πάρης αργότερα θα σας μιλήσει για το θέμα αυτό. Πάντως αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να καθορίσει τα πολιτικά κριτήρια αυτού του συστήματος αλλά και τα στρατιωτικά κριτήρια ενός τέτοιου συστήματος. Και μετά θα δούμε πώς μια και το διάστημα εκφύσεως έχει δραστηριότητες διτής χρήσης, θα δούμε πώς θα διαμορφώσουμε ένα σύστημα που θα ανταποκρίνεται όχι μόνο στις ε, πολιτικές μας ε, απαιτήσει και φιλοδοξίες, αλλά και στις ε, στρατιωτικές απαιτήσει μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, του ΕΝΤΑ και των κρατών μελών. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα είναι πραγματικό σύστημα dual use, διπλής χρήσης, πολιτικό και στρατιωτικό. Έχουμε φυσικά, είπαμε αυτό το θέμα, είναι, αφορά την ασφάλεια του διαστήματος. Έχουμε όμως και ένα δεύτερο σκέλος που αφορά τη χρήση της τεχνολογίας, είτε το GMS, e είτε το Γαλιλαίο, είτε το πρόγραμμα γεωσκόπηση είτε το Γαλιλαίο. Αυτή η τεχνολογία διτής χρήσης ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, αλλά πώς θα εξασφαλίσουμε την εξυπηρέτηση και ε, πολιτικών ασφάλειας με το σύστημα αυτό. Για το σύστημα γεωσκόπησης, το GMS, e θέλουμε να δούμε πώς, με ποιο τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε το GMS e και επαναλαμβάνω, το GMS e δεν είναι μόνο σύστημα γεωσκόπησης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος, έχει και το, εκτός από το environment, το e, έχει και το S που είναι παρακολούθηση και της ασφάλειας αυτό το γεωσκοπικό σύστημα. Οπότε προσπαθούμε να αναπτύξουμε και το σκέλος ασφάλειας του GMS, παρακολούθηση περιβάλλοντος και ασφάλειας. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να καθορίσουμε κάποιες εφαρμογές, να προσδιορίσουμε κάποιες εφαρμογές για τη χρήση του GMES στα θέματα επιτήρησης συνόρων και εκεί συνεργαζόμαστε και με άλλες μονάδες και διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαίους εταίρους για να καταλήξουμε σε ένα κόνσεπτ και σε μια πολιτική για το GMES για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε το GMES. Επίσης θέλουμε να προσδιορίσουμε κάποια κριτήρια για να δούμε πώς μπορεί να στηρίξει το GMES και τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένας τρίτος τομέας είναι πώς μπορεί να βοηθήσει το GMES για την παρακολούθηση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Δεν είναι μυστικό, το έχει δηλώσει από την αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι ένα σύστημα όπως το Γαλιλαίο μπορεί να έχει και στρατιωτική χρήση. Παρόλο που είναι καταρχήν σύστημα ελέγχου μη στρατιωτικό. Αυτή τη στιγμή πάντως γίνονται συζητήσεις για το πώς το PRS, το Public Restricted Services του Γαλιλαίου μπορεί να αξιοποιηθεί και για δραστηριότητες ασφάλειας. Βέβαια, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της ε, άσκησης των αρμοδιοτήτων μας, γιατί το, η συνθήκη της Λισαβόνας μας βοηθάει από νομική άποψη. Καταργήθηκαν οι πυλώνες, θεωρητικά τουλάχιστον. Οπότε έχει ξεκινήσει ένας διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και θα δούμε πώς πέρα από τα βήματα που σας ανέφερα εγώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερες συνεργασίες για να αξιοποιήσουμε τις διαστημικές μας δραστηριότητες και για πολιτικούς λόγους, μη στρατιωτικούς, αλλά και για θέματα ασφάλειας και άμυνας. προσπαθούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να καταλήξουμε και σε συμφωνίες ε, για κοινέ δραστηριότητε. Βέβαια, πολλά στοιχεία, ιδιαίτερα του διαστήματος, ό,τι αφορά δραστηριότητες ασφάλειας, ε, εναπόκεινται στα κράτη-μέλη. Και πολλές φορές υπάγονται σε στρατιωτικά ζητήματα, σε στρατιωτικό έλεγχο ή στον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας. Οπότε, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε πραγματικές συνέργειες μεταξύ μη στρατιωτικού και στρατιωτικού κλάδου, φυσικά θα προσκορούσουμε σε κάποιους περιορισμούς και επιφυλακτικότητα από άποψη των στρατιωτικών. Γιατί χρειάζεται εμπιστοσύνη και χρειάζεται ανάπτυξη του διαλόγου για να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε και τα δύο σκέλη, το στρατιωτικό και το μη στρατιωτικό, για να συνεργαστούμε, να ανταλλάξουμε πληροφορίες ή και δεδομένα και από, και από τα δύο σκέλη. Και για τον προβληματισμό αυτό σκεφτόμαστε ότι ε, ναι, το χρειαζόμαστε και πρέπει να δούμε τι απαιτείται για να το συνεχίσουμε αυτό στο μέλλον, για τον διάλογο με τα κράτη-μέλη, ποιοι είναι οι συνομιλητές τους οποίους πρέπει να συμπεριλάβουμε. Αυτός ο προβληματισμός αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή και όπως σας είπα από νομική άποψη, ναι, η συνθήκη με τα άρθρα και τις αλλαγές που εισήγαγε τουλάχιστον θεωρητικά διευκόλυνε τα πράγματα. Αλλά πάντοτε υπάρχουν και ε, τα πρακτικά ζητήματα, πώς να οργανωθεί αυτός ο χώρος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών, πώς θα οργανωθεί μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ δύο των τομέων σε επίπεδο εφαρμογών. Πέρα από αυτό, όπως είπα, τα επόμενα στάδια, έτσι πιο συγκεκριμένα, ποια είναι. Σε γενικές γραμμές, όπως ανέφερα και νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή ε, εξετάζει ποιους, ποιες εμπλεκόμενες πλευρές, ποια κράτη-μέλη, ποιοι Ευρωπαίοι εταίροι ε, πρέπει να συμμετέχουν και ποια πρέπει να είναι η στρατηγική της Ευρώπης για το διάστημα στο μέλλον. Υπάρχει φυσικά και η προετοιμασία του νέου οικονομικού πλαισίου, του επόμενου οικονομικού πλαισίου, το οποίο θα μπει στην του, στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του χρόνου θέλουμε μετά από τις συζητήσεις ε, που θα κάνουμε με, με τα άλλα όργανα, με τους άλλους θεσμούς, με τα κράτη-μέλη, με τις εμπλεκόμενες πλευρές, θέλουμε να φέρουμε συγκεκριμένες ιδέες για κάποιες προγρα... ή κάποιες προγραμματικές προτάσεις για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, εφόσον έχουμε την αρμοδιότητα και εφόσον έχουμε φιλοδοξίες στον τομέα για το μέλλον, για τα επόμενα 7 με 10 χρόνια πρέπει επίσης να αποκτήσουμε και τα μέσα και τα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να εφαρμόσουμε αυτές τις ιδέες. Θέλουμε λοιπόν να εκφράσουμε αυτές τις ιδέες με προγραμματικές προτάσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν περίπου στα μέσα του επόμενου έτους θα έλεγα. Πάντοτε φυσικά σύμφωνα με το γενικό προγραμματισμό των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων για τον συνολικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω πια εδώ και να δώσω λίγο χρόνο και στους συναδέλφους την, από, την ΕΣΑ και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας να μας πούν και τη δική τους άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, η κυρία Ναζά από τον από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, χωρίς να θέλω να υπησέλθω στο περιεχόμενο της ομιλίας σας. Ε, νομίζω ότι ήταν, ε, θέλουμε κάτι πολύ έτσι διδακτικό και μεστό νοήματος. Να μας πείτε τι ακριβώς, πώς ακριβώς εμπλέκεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος σε αυτό το θέμα. Oui, bon. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το, καλό, το πλεονέκτημα με το ότι μιλάω μετά από τη συνάδελφο είναι ότι κάλυψε πάρα πολλά θέματα και έτσι εγώ θα μπορέσω τώρα να επικεντρώσω την προσοχή μου στην προστιθέμενη αξία της ε, ΕΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, σε αυτό το νέο πλαίσιο, το διαστημικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Εν συντομία... Εν συντομία λοιπόν, η Σίλβια το είπε ήδη. Το διάστημα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που εντάσσεται σε πολλές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως πολιτικές που έχουν χαρακτήρα άμυνας και ασφάλειας, αλλά και γενικότερα έχουμε τη γενική επιτήρηση του περιβάλλοντος, της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της κοινωνίας της πληροφορίας κτλ. Με ρωτήσ, μου ζητήσατε να γίνω λίγο πιο ειδική και να μιλήσω για τον ιδιαίτερο ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Ο ΕΟΔ λοιπόν είναι μια διακυβερνητική, ένας διακυβερνητικός φορέας, ο οποίος ιδρύθηκε το 1975 από τα ευρωπαϊκά κράτη, έχει 18 μέλη αυτή τη στιγμή, ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία σε γενικές γραμμές είναι τα ίδια μέλη με την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την διεύρυνσή της, μόνο που υπάρχει ακόμα και η Νορβηγία και η Ελβετία. Δεν έχουν γίνει μέλη μας ε, ακόμα όλα τα καινούργια μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδιαφέρον έχει δείξει η Ρουμανία, η Τσεχία, η Ρουμανία μάλιστα θα γίνει μέλος πάρα πολύ σύντομα και θα διευρυνθούμε τα επόμενα χρόνια. Ε, και στο τέλος θα συμπεριλαμβάνουμε και εμείς τα ίδια κράτη-μέλη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα έχουμε συμφωνίες με όλα σχεδόν τα κράτη. Έχουμε περίπου 2.000 άτομα προσωπικό ε, σε διάφορους φορείς διάσπαρτους στην Ευρώπη. Έχουμε έναν προϋπολογισμό 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ Κάτι σημαντικό που πρέπει νομίζω να εξηγήσω είναι ότι ο ΕΟΔ καλύπτει όλες τις διασταμικές δραστηριότητες. Αντίθετα με τη μεγάλη του αδερφή την NASA, ε, η οποία εστιάζεται στους τομείς της επιστήμης και, του, και της, της ενίκησης του διαστήματος. Ο ΕΟΔ αντίθετα καλύπτει όλους τους τομείς, τις εφαρμογές, την τεχνολογία, την επιστήμη, τους πυράβλους. Επίσης είναι ε, Προφανώς όμως οι επενδύσεις μας είναι χαμηλότερες από ό,τι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, ε σημειώθηκαν μεγάλες επιτυχίες. Έχουμε αναπτύξει και εκτοξεύσει καμιά εξενταριά δορυφόρους. Επίσης κάνουμε, οι δορυφόροι αυτοί έχουν τεχνολογικό, επιστημονομικό περιεχόμενο επιτήρησης του περιβάλλοντος. Έχουμε δύο πιλωτικά προγράμματα για τον Γαλιλαίο. Ε, μια δραστηριότητα λοιπόν που καλύπτει όλες τις πτυχές του διαστήματος. Θα ήθελα ίσως ε, εντάχει να πω ε, τι κάνει, πώς λειτουργεί αυτή η διακυβερνητική οργάνωση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους εκπροσώπους των κρατών μελών ε, που συμμετέχουν ε, σε ένα συμβούλιο. Έχουμε δύο τύπους προγραμμάτων. Υποχρεωτικά προγράμματα, το περίπου το 15% των προγραμμάτων μας και αφορούν τεχνολογικά και επιστημονικά προγράμματα και στη συνέχεια έχουμε τα προαιρετικά προγράμματα ε, εφαρμογές, ε, εκτοξεύσεις, ε, εφαρμογές σε όλους τους τομείς, παρατηρητήρια, τηλεπικοινωνίες, πλοήγηση και το, τα προγράμματα αυτά τα κράτη επιλέγουν σε ποια προγράμματα θα συμμετέχουν και ποιο θα είναι το ύψος της συμμετοχής τους. Ε, είναι λοιπόν ένας οργανισμός αρκετά ευέλικτος αφού τα κράτη μπορούν να επιλέξουν αν θα συμμετάσχουν ή όχι στα προγράμματα ανάλογα με τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντά τους γιατί ένας άλλος κανόνας του ΕΟΔ είναι η βιομηχανική του πολιτική η οποία βασίζεται πάνω απ' όλα στον ανταγωνισμό αλλά η οποία στοχεύει επίσης και στην εξασφάλιση μιας ισόρροπη ε, συμμετοχής και εφαρμογή των κρατών μελών, μια συμμετοχής που είναι ανάλογη της συνεισφορά τους. Υπάρχει ο κοινός κανόνας που είναι το γεωγραφικό ρετούρ που σύμφωνα με το οποίο είναι ένα είδος απόδοση, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη εποφελούνταν στο βαθμό που συνεισφέρουν οικονομικά στην ανάπτυξη των προγραμμάτων. Ε, έχει περάσει αρκετό καιρός που εργαζόμαστε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα Γαλιλαίο και το ΖΕΜΕΣ είναι προγράμματα τα οποία είχαν τεθεί σε εφαρμογή πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας, οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη είχε έναν ενεργό ρόλο στο διάστημα. Απλώς με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας δίδεται και ένα πολιτικό βάρος σε αυτή τη διαστημική δραστηριότητα. Η Σίλβια το ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται από, μια συμφωνία πλαίσιο, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 2004. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής συστάθηκε το Συμβούλιο Διαστήματος, που είναι κοινό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΔ, και που συνέρχεται τακτικά. Από το 2004 συνήλθε έξι φορές. Ε, ε, ε, θα υπάρξει η έβδομη συνεδρίαση στις 25 Νοεμβρίου που μας έρχεται. Σε μία τέτοια συνεδρίαση το 2007 τα 29 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΔ υιοθέτησαν ένα ψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική ε, το 2007 λοιπόν, αυτά τα 29 χρόνια, ανέλαβαν μια ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική η οποία καθόριζε τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους για το διάστημα ε, την ανάπτυξη διαστημικών εφαρμογών στην υπηρεσία της, πολιτικής, της ευρωπαϊκής πολιτικής και του ευρωπαίου πολίτη, την ανάγκη να καλυφθεί η ασφάλεια και η άμυνα και από τις διαστημικές πτυχές, ε, η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία για τον διαστημικό κλάδο, η συμβολή της κοινωνίας της πληροφορίας και η έννοια που είναι πολύ σημαντική νομίζω ιδίω για τη δική σας επιτροπή, η άποψη μάλλον ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει μια εγγυημένη πρόσβαση ε, στα συστήματα και στις ικανότητες χωρίς να παρεμποδίζεται από τεχνολογικά εμπόδια, έτσι ώστε να μπορεί να έχει μια ισορροπημένη πολιτική. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν θα επανέλθω σε όσα υπόθηκαν. Υπάρχει αυτή η συμφωνία πλαίσιο που ισχύει μέχρι το 2012 και στη συνέχεια θα δούμε αν πρέπει να την επικαιροποιήσουμε ή να την παρατείνουμε ή να την προσαρμόσουμε. Υπάρχει λοιπόν το Συμβούλιο για το διάστημα που ιδρύθηκε το 2004, το πλαίσιο συνεργασίας με τα κράτη-μέλη κτλ. Η Σίλβια επίσης ανέφερε, πέρα από αυτή τη συμφωνία πλαίσιο, έχουμε τον λεγόμενο διαρθρωτικό ή δομικό διάλογο για το διάστημα και την ασφάλεια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΤΕα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τον ΕΟΔ και όλοι μαζί συζητούν όλα αυτά τα θέματα ασφάλειας και διαστήματος. Και τέλος, για να, να είναι ολοκληρωμένη η παρουσίασή μου, πρέπει επίσης να πω ότι υπάρχει μια καινούργια συνεργασία με την DEA ε, για τις τεχνικές. Είναι μια διοικητική δομή η οποία θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε και να προάγουμε ακόμα περισσότερο αυτήν τη συνεργασία. Ίσως λοιπόν για να μιλήσουμε επίσης για το θέμα που σας ενδιαφέρει πιο ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Επιτροπής αυτής, το θέμα της ασφάλειας, συχνά λέγεται ότι δεν υπάρχει κάποιος οργανισμός που να εφαρμόζει προγράμματα ασφάλειας. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Η συνθήκη δεν λέει, ε, ε, ορίζει ότι ο ΕΟΔ είναι ένας πολιτικός οργανισμός και διεξάγει δραστηριότητες όμως με αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς μη επιθετικούς, μη επεμβατικούς όπως καθορίζονται από το καταστατικό του ΟΗΕ. Ε, μπορούν λοιπόν ο οργανισμός αυτός να εφαρμόσει προγράμματα ασφάλειας και άμυνας αρκεί να είναι πολιτικής φύσεως, να χρηματοδοτούνται από τον πολιτικό προϋπολογισμό και ε, από εδώ και στο εξής αναπτύσσουμε τεχνολογίες ε, τέτοιας χρήσης ε, Άμυνας και Ασφάλειας. Η Σίλβια ανέφερε την εποπτεία του διαστήματος. Υπάρχει ένα κονδύλιο που δίδεται από τα κράτη-μέλη και προέρχεται από το Υπουργείο Άμυνας. Λίγο-λίγο ε, λοιπόν, γλυκά-γλυκά ε, μπαίνουμε και εμείς σε αυτόν τον τομέα άμυνας και ασφάλειας. Έχουμε και τον, ε, τη συμμετοχή μας σε αυτόν τον δομικό διάλογο που δημιουργεί το πλαίσιο και συγκεκριμενοποιεί τα βήματα προόδου στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η πρόκληση σήμερα είναι φυσικά η επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας που για εμάς είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να ενισχύσουμε την πολιτική ορατότητα του διαστήματος και να θέσουμε το διάστημα στην υπηρεσία της πολιτικής και συγκεκριμένα της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Το παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η συνθήκη αφού για πρώτη φορά κάνει λόγο για το διάστημα. Πρώτη φορά μια Ευρωπαϊκή Συνθήκη κάνει λόγο για το διάστημα σε συνδυασμό με την άμυνα ε, και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ε, το βλέπουμε ως κάτι πάρα πολύ χρήσιμο για να πολλαπλασιάσουμε και να εμβαθύνουμε τις δραστηριότητες μας στον τομέα. Ένα άλλο σημείο που έχει ενδιαφέρον για μας είναι η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που για μας θα γίνει ένα μέσο κεντρικής σημασίας και που πραγματικά θα χρειαστεί και ένα διαστημικό εργαλείο. Προσπαθούμε ακριβώς να δημιουργήσουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Όπως είπε και η Σίλβια, υπάρχουν προγράμματα που παρότι είναι πολιτικής φύσεως μπορούν ε, να έχουν διτή χρησιμότητα, στρατιωτική χρησιμότητα, συγκεκριμένα το ΖΕΜΕΣ και το Γαλιλαίο. Άλλο πάλι πρόγραμμα ε, που αναπτύσσουμε και που έχει ε, έντονο βάρος για το στρατιωτικό κομμάτι είναι ένα πρόγραμμα για την μείωση του χρόνου απόκτησης δεδομένων και διάδοσης δεδομένων κατά πολλές ώρες σε 5-6 λεπτά, 1 τέταρτο κατελάχιστον. Καταλαβαίνετε ότι ένα σύστημα διαβίβασης δεδομένων ταχύ επιτρέπει μια πολύ καλύτερη πρόσβαση στα στοιχεία και αυτό από πλευράς άμυνας και ασφάλειας είναι κέριο. Η Σίλβια μίλησε επίσης και για ένα άλλο πρόγραμμα, ίσως και ο Πάρης να μιλήσει γι' αυτό. Είναι το σύστημα διαστημικής επιτήρησης παρακολούθησης του διαστήματος. Ε, όπως ξέρετε η πολίτες ε, έχουν ανάγκη από αυτές τις διαστημικές ε, δομές προστασίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι που απειλούν τις υπηρεσίες μας. Ε, υπάρχουν τα λεγόμενα διαστημικά σκουπίδια, απορρίμματα. Υπάρχει το πρόβλημα αποφυγής των συγκρούσεων. Υπάρχει το πρόβλημα προστασίας από τους αστεροειδείς αλλά και από τις ηλιακές θύελες. Ο στόχος λοιπόν του προγράμματος αυτού ε, από το 2012 θα είναι σημαντική χρονιά ε, γι' αυτό, γιατί θα περάσουμε στην επιχειρησιακή φάση του προγράμματος, το οποίο αυτή τη, προς το παρόν βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας. Είναι όμω ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα όπου η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι τόσο η εφαρμογή της, των διαστημικών εφαρμογών, αλλά το στήσιμο μια διαστημική ε, αρχιτεκτονική που συνδυάζει τα χερσαία με τα διαστημικά εργαλεία και μέσα, γιατί υπάρχουν. Ε, υπάρχουν ήδη για αρκετά χρόνια σε εθνικό επίπεδο. Ο στόχος λοιπόν είναι να συνδυαστούν επιτυχώς οι χερσαίες και διαστημικές υποδομές. Ένα τελικό σημείο, η ε, διαχείριση των κρίσεων. Στον ΕΟΔ είμαστε πεπισμένοι ότι τα διαστημικά μέσα έχουν πολύ μεγάλη χρησιμότητα για τη διαχείριση των κρίσεων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, ε, συναντούμε κάποιες αντιστάσεις βέβαια, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι στον τομέα αυτό πραγματικά θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε πολύ περισσότερο. Θέλω να αναφέρω ήδη ότι υπάρχει μια χάρτα, μια διεθνής χάρτα για μείζονες ε, καταστροφές με στόχο την πολιτική προστασία με την παροχή διαστημικών εικόνων που καταγράφουν οι δορυφόροι από τις διάφορους διαστημικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο. Ε, να σας πω ότι η Γαλλική Διαστημική Υπηρεσία ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη αυτής της χάρτας. Είναι μια χάρτα που λειτουργεί πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ αποτελεσματική, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε και περισσότερο στον τομέα αυτό. Εξού και η πρωτοβουλία μας να σκεφτούμε τη δημιουργία μιας υποδομής ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για την αντιμετώπιση των κρίσεων, είτε πρόκειται για φυσικές θεομηνίες, είτε για παρεμβάσεις ε, σε καιρό ειρήνης. Όλο το φάσμα των κρίσεων λοιπόν πιστεύουμε ότι μπορούμε να το στηρίξουμε και να διαχειριστούμε καλύτερα με διαστημικά μέσα και ακριβώς προβληματιζόμαστε πάνω σε αυτό. Και με τον συνάδελφο βέβαια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Ε, και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας, ε, ένα μεγάλο λιθαράκι και να βοηθήσουμε και εμείς την οικοδόμηση αυτής της Ευρώπης ως, πολιτική δύναμη, ως πολιτικής δύναμης. Η Σίλβια, όπως είπε και η Σίλβια, πολλά πράγματα έχουν γίνει μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Έχουμε πλέον το Συμβούλιο Διαστήματος, το οποίο θα συνέλθει τον επόμενο μήνα και που θα είναι μια ευκαιρία ενίσχυσης και πρόοδου πάνω στο θέμα αυτό. Το 2011 θα έχουμε την διοικητική συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας που θα τεθεί σε ισχύ. Το 2012 θα είναι η χρονιά που ε, θα εδρεώσουμε το πρόγραμμα επιτήρησης στο διάστημα. Το 2012 θα έχουμε και μια νέα διυπουργική συνάντηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για τον προϋπολογισμό μας και όπως είπε και η Σίλβια πιστεύω ότι στη διάρκεια των ε, χρόνων αυτών θα προετοιμαστεί και το δημοσιονομικό, το χρηματοδοτικό πλαίσιο ε, της Ευρώπης το οποίο θα συγκεκριμενοποιήσει τις φιλοδοξίες της Ευρώπης για το διάστημα. Νομίζω λοιπόν ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι κέρια για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα. Σας ευχαριστώ και τέλος ο κύριος Πάρης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Θα μας μιλήσει για τις ε, δορυφορικές επικοινωνίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας ε, ευχαριστήσω που καλέσατε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας ε, και μας δώσει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα διαστήματος, ασφάλειας και άμυνας κυρίως μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας που αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χαράξει τη δική της πολιτική διαστήματος και να ε, προάγει την εφαρμογή των συναφών πολιτικών, οι οποίες πολιτικές επελαμβάνουν την κοινή ε, πολιτική άμυνας και ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την υπεραξία του διαστήματος ε, κυρίως στον ε, σχεδιασμό και τη διαχείριση των κρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μας δίνει πλέον μια νέα διάσταση σε όλο αυτό το θέμα να υπάρχει μια πιο ε, εκτεταμένη προσέγγιση. Όσον αφορά λοιπόν τον δικό μα τον οργανισμό, ο συνθήκη τη Λισαβόνα μας δίνει συγκεκριμένε αρμοδιότητες στην άμυνα, στον προγραμματισμό, στην έρευνα, να εντοπίσουμε ε, τις λειτουργικές ανάγκες, να προάγουμε τα μέτρα για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες αυτές και να συμβάλλουμε στο να ενισχυθεί η ε, τεχνολογική βάση του τομέα τη Άμυνα. Άρα δηλαδή ε, υπάρχουν αυτές οι αρμοδιότητες για τον φορέα μας και αυτό προφανώς περιλαμβάνει και το διάστημα όπου έχουμε συνάψει στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με, ε, με τον Οργανισμό Διαστήματος και με το Συμβούλιο μέσα από το διαρθρωμένο διάλογο που έχει λάβει η χώρα τα τελευταία χρόνια για την ασφάλεια του διαστήματος. Θα αναφερθώ λοιπόν σήμερα σε δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα στο θέμα του διαστήματος ε, μέσα από μία προσέγγιση των δυνατοτήτων που υπάρχουν και δεύτερον στις ευκαιρίες που προσφέρει έτσι ώστε να ενισχυθεί η στρατιωτική και η πολιτική συνεργασία, ένα θέμα που είναι πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη του φορέα μας, όπως ανέφεραν και οι προλαλήσαντες. Ε, ο Οργανισμός Άμυνας έχει και αυτός κάποιες αρμοδιότητες. Το θέμα λοιπόν του διαστήματος πρέπει να εξαρθεί κάτω από το πρίσμα των δυνατοτήτων, δηλαδή δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε μια γκάμα μέτρων και πρωτοβουλειών έτσι ώστε να προκαλέσουμε το ε, προσδοκόμενο αποτέλεσμα το οποίο θα πρέπει να λάβει χώρα σε όλα τα επίπεδα, το στρατηγικό, ε, το επιχειρησιακό ε, και ε, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επίσης. Αυτές λοιπόν οι δυνατότητες αφορούν όχι μόνο συστήματα αλλά αφορούν και συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αφορούν οργανισμούς, ε, τη διακυβέρνηση και την διαχείριση πληροφοριών. Και αυτό περιλαμβάνει και το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και την ασφάλεια ε, δικτύων πληροφοριών γενικότερα. Μιλάμε λοιπόν για συστήματα τα οποία συμβάλλουν σημαντικά σε τομείς όπως είναι η αναγνώριση και η παρακολούθηση. Άισα που ε, ασχολείται με το διάστημα ανακοινώσεις ε, SATCOM ε, Satellite Communication ανακοινώσεις για το διάστημα επίσης πρέπει να υπάρχει και περαιτέρω χρήση συγκεκριμένων πληροφοριών έτσι ώστε να υπάρχουν στοιχεία για την τοποθέτηση και την πλοήγηση. Εδώ γίνεται ε, σχεδιασμός με το Γαλιλαίο. Αυτό που ενδιαφέρει να υπάρχει και πληροφορία σχετικά με, το μετρολογικό. Εμείς λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι το κέντρο, να το διάστημα να μην ε, αφορά μόνο αυτό αλλά να χρησιμοποιήσουμε και τις απαραίτητες πληροφορίες για όσους χρησιμοποιούν το διάστημα. Και το πιο σημαντικό κριτήριο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ευελιξία στη χρήση, αντίδραση, δυνατότητα αντίδρασης, ασφάλεια και παροχή υπηρεσιών, ε, κόστος ε, και διάρκεια παροχής υπηρεσιών. Το δεύτερο σκέλος ε, αφορά στην διτή διάσταση ε, του διαστήματος, το οποίο διάστημα από τη φύση του έχει ένα διτό χαρακτήρα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι πώς μπορεί κανείς να ανταποκριθεί στις ε, ανάγκες αναγνώρισης όσον αφορά στο διάστημα. Μέχρι τώρα τα περισσότερα προγράμματα του διαστήματος ήταν είτε στρατιωτικά συστήματα είτε μη στρατιωτικά, πολιτικά. Ακόμα και υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Ο χώρος του διαστήματος ε, μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα εργαλείο διτό το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες και των δύο τομέων χάρη της σύγκλησης των ε, αναγκών ε, γιατί ε, λαμβάνουν χώρα πολλές φορές και στρατιωτικές και μη στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τηλεπικοινωνιακά, πλοήγηση σε ένα ασφαλές περιβάλλον, δυνατότητα αντίδρασης. Αυτά θα, εκεί θα υπάρχει πάντα ανάγκη να υπάρχει έρευνα και σε στρατιωτικό και σε μη στρατιωτικό επίπεδο Πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να γίνει εξωτερική ανάθεση ε, των ερευνών όπου εμπορικοί οργανισμοί θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ε, λύσεις ε, για τους χρήστες συστημάτων άμυνας. Εδώ ε, το SATCOM, χωρές SATCOM της ε, δορυφορικής επικοινωνίας είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα εξαρτώμεθα από εμπορική παροχή πληροφοριών και παράλληλα υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα που μπαίνει για την Ευρώπη δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να έχει εγγυημένη πρόσβαση σε καθοριστικά ε, δίκτυα και συνδέγους επικοινωνίας όπως είναι αυτά για το στρατιωτικό τομέα εδώ ξεκινάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το μηδέν και αυτό ισχύει και για την παρατήρηση της γης ε, όπου ε, δίδονται οι πληροφορίες από ε, providers εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλουμε λοιπόν να βασιζόμαστε σε πληροφορίες που αφορούν μόνο την Ευρώπη και προσφέρονται από την Ευρώπη και τα κράτη-μέλη, είναι πολύ σημαντικό όλο και περισσότερο με διαρθρωμένο διάλογο να αναπτύξουμε τις δυνατότητες. Πρέπει να αναλύσουμε πολύ προσεκτικά τις ανάγκες ε, που υπάρχουν ε, στον στρατιωτικό και στον πολιτικό τομέα, έτσι ώστε να μπορούμε να βασιστούμε σε ε, ένα, μια σειρά αναγκών όπου να μπορεί να ανταποκριθεί αυτό το διτό σύστημα. Και η πρώτη πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τέτοιο πείραμα στο SSA ε, που έχει ως στόχο να έχουμε ένα σύστημα διτό που θα εξυπηρετεί τόσο τον αισθητικό όσο και το μη στρατιωτικό τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να σας προσφέρω και ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα ε, του τι έχουμε κάνει εμείς μέχρι σήμερα. Όσον αφορά τον συντονισμό των επενδύσεων σε ε, έρευνα και τεχνολογία για το διάστημα, εδώ λαμβάνονται υπόψη δύο στοιχεία. Πρώτον, όσον αφορά στη διαθεσιμότητα κέρυας διαστημικής τεχνολογίας για εξωτερικές πηγές, ΙΖΑ, Κομισιόν, EDA, όλοι αυτοί έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να εντοπίσουν σημαντικούς τομείς της τεχνολογίας και για να μπορέσουν να εναρμονίσουν τους κανόνες εφαρμογής. Δεύτερον, συντονισμένες αποστολές επίδειξης ανάμεσα στην EDA και την ΙΖΑ, ανάμεσα σε αυτούς φορείς έχουν ξεκινήσει ως ε, πρώτες πειραματικές περιπτώσεις ε, στον τομέα της ε, δορυφορικής επικοινωνίας και αυτό για να υπάρχει μια παγκόσμια χρήση. Να υπάρχει λοιπόν πιο συστηματική προσέγγιση. Για να το πετύχουμε αυτό ξεκινήσαμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ίζα και με το Συμβούλιο το ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας που έχει ως στόχο μεγαλύτερη συνεργασία, συμπληρωματικότητα ανάμεσα στην αστική ασφάλεια, το διάστημα και την έρευνα που έχει σχέση με το διάστημα. Και αυτή τη στιγμή ερευνούμε συγκεκριμένους τομείς, έχουμε το CBRN, αλλά επίσης ε, και αυτό που έχει μεγαλύτερη σχέση με το διάστημα, το US και τομείς όπου μπορούμε πράγματι να συνεργαστούμε. Το δεύτερο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ο συντονισμός ε, ε, σχετικά με τον ορισμό των αναγκών ε, και θα ήθελα να αναφέρω τρία παραδείγματα από αυτού. Πρώτον, η ομάδα που να αφορά τη συνεργασία της στρατιωτική για παρατήρηση στη γη έχουμε δύο προγράμματα παρατήρησης ε, τα οποία ε, δρομολογήθηκαν ξεχωριστά το καθένα από αυτά ε, αντίστοιχα στο στρατιωτικό και τον μη στρατιωτικό τομέα. Υπάρχουν λόγοι για τέτοιου της προσέγγιση αλλά καθίστατε όλο και περισσότερο σαφές ότι μπορεί κανείς να αναζητήσει τη συνεργασία ανάμεσα αυτούς τους δύο τομείς. Μπορούν και οι στρατιωτικοί να χρησιμοποιούν πολιτικά συστήματα και τα νάπαλιν. Βέβαια αυτό είναι μια δύσκολη διαδικασία και θα πρέπει να προχωρήσει μπορούμε βέβαια να αναζητήσουμε και δυνατές συνεργασίες απ' έξω όταν θα εξετάσουμε τις δυνατότητες της επόμενης γενιάς. Οι μελλοντικέ ε, εξελίξεις όσον αφορά την διάσταση ασφαλείας του GMS μπορούν επίσης να επηρεαστούν από, αυτές τις, ε, τους, από αυτούς τους προβληματισμούς. Όσον αφορά την ε, ευαισθητοποίηση για το διάστημα SSS με το οποίο ασχολούμαι τώρα. Ξεκινήσαμε τον ορισμό ε, των αναγκών ε, που ε, προχωράει παράλληλα με το EDA και την ΙΖΕ και αφορά και σε ανάγκες στρατιωτικών χρηστών και μη στρατιωτικών. Πολλές από τις ανάγκες αυτές είναι συμπληρωματικές για να μην μπούμε ταυτόσιμες. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που αφορούν την άμυνα, παραδείγματος χάνει την ανάγκη να υπάρχει αναγνώριση στο διάστημα. Και αυτό αφορά εικόνες που έχουν έχουν σχέση με το διάστημα αλλά και με τη γη. Αυτό που πράγματι υπάρχει είναι ότι υπάρχει δυτή χρήση των διεθνών συμβάσεων που σημαίνει οι ε, πολιτικοί χρήστες πρέπει να δειχθούν ε, την αυστηρή χρήση των ε, αναγκών όσον αφορά τις κυβερνήσεις και την πολιτική για τα δεδομένα. Επιπλέον όσον αφορά τις πληροφορίες ε, και την αναγνώριση ε, και σε αυτόν τον τομέα η συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους είναι καθαριστικής σημασίας έτσι ώστε να υπάρχει το απαραίτητο μείγμα ανάμεσα σε ε, πόρους που έχουν σχέση με το διάστημα και άλλους εκτός αυτού. Αφού λοιπόν θα υπάρχουν ε, κοινοί στόχοι, η EDA θα ε, εξετάσει σε μία περαιτέρω μελέτη αρχιτεκτονικές δυνατότητες, ας τις αποκαλέσουμε έτσι, ε, πακέτων που θα αφορούν λειτουργίες με την βέλτιστη σχέση κόστους. Όσον αφορά και αυτή είναι, αυτό είναι το τελευταίο μου παράδειγμα, επίσης ένα πρόγραμμα με το οποίο ασχολούμαι, όσον αφορά στην έρευνα για λύσεις αποτελεσματικές από πλευράς κόστους, η DS δρομολόγησε ένα πρόγραμμα που φέρει τον τίτλο ESCPC, το οποίο θα μπορεί να προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη τηλεπικοινωνικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικούς όρους, επιτρέποντάς τους ε, να ε, εντάξουν ε, και την ευρωπαϊκή ζήτηση λόγω της κεντρικής παροχής. Αυτό λοιπόν είναι ένα συγκεκριμένο εργαλείο, τουλάχιστον ανοίγει το δρόμο, που μπορεί να επεκταθεί το όλο θέμα προς την παρατήρηση ή ε, προς ε, κυβερνητικές, ε, δορυφορική, κυβερνητική δορυφορική επικοινωνία. Ίσως ε, να χρειαζόμαστε ε, κάποια ειδική στρατηγική με το διάστημα, αλλά το διάστημα πρέπει να ενταχθεί σε, άλλες, σε άλλα προγράμματα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η ε, ευρύτερη στρατιωτική και πολιτική διάσταση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματο, το Συμβούλιο και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα πρέπει να συνεχίσουν το διάλογο για θέματα ασφάλεια και να αυξήσουν το συντονισμό, να τον προάγουν περαιτέρω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια η οποία στοχεύει στο να προστατέψει και να διασφαλίσει την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Euh, σας ευχαριστούμε για την διεξοδικότητα αυτή παρουσίαση. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις προς την κυρία Ναζά πολύ συγκεκριμένες. Αναφερθήκατε στο Συμβούλιο Διαστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται αυτό το Συμβούλιο Διαστήματος. Αναφερθήκατε σε 29 μέλη αυτού του Συμβουλίου. Δηλαδή 27 από τις ευρωπαϊκές χώρες, άρα δύο μη ευρωπαϊκές ε, χώρες, μη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι δύο εξοκοινωτικές χώρες που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Διαστήματος. Επίσης μιλήσατε για τη σχέση με τις τρίτες χώρες και κυρίως τις αναδυόμενες, ε, ραγδαία αναδυόμενες ε, οικονομίες και στον ε, διαστημικό κλάδο, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία. Τι γίνεται με αυτές, ποια είναι η συνεργασία με τις χώρες αυτές. Επίσης, στο ΝΑΤΟ γίνεται λόγους ε, για την αντιπυραυλική άμυνα. Τι γίνεται με τα διαστημικά προγράμματα έγκυρης προειδοποίησης, γιατί μερικές χώρες ασχολούνται μεμονωμένα με αυτό το θέμα. Μπορούμε στα υπερεθνικά τέτοια όργανα και οργανισμούς να μεταθέσουμε αυτή τη συζήτηση για την αντιπυραυλική άμυνα, γιατί πολύ λόγος γίνεται το τελευταίο καιρό. Κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τους ε, τρεις εισηγητές ε, για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις που ακούσαμε. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε συστήσει πλέον ε, αρκετούς οργανισμούς ε, που έχουν συγκεντρώσει ειδική τεχνογνωσία και τώρα πλέον πρέπει να επιδείξουμε πολιτική βούληση για να εφαρμόσουμε όλα αυτά που έχουμε κατακτήσει. Ε, εσείς μεταξύ άλλων μιλήσατε για την χρήση μορφών συνεργασίας, συνέργειες, συνεργασία στρατιωτικής και μη στρατιωτικής μορφής να υπάρξει λοιπόν μια ε, σύγκληση των ε, αναγκών η οποία μπορεί να προκύψει όταν ε, υπάρξουν συνεργασίες ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα που προέκυψε για μένα. Πολύ συγκεκριμένα, στο τέλος της παρέμβασής σας είπατε ότι το Συμβούλιο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας πρέπει να παραμείνουν σε διάλογο σχετικά με τις ανάγκες, με το τι είναι απαραίτητο. Αυτό βέβαια με εκπλήσει λιγάκι γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας είναι ένας οργανισμός που κατ' ουσίαν δέχεται εντολές. Δηλαδή ε, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ε, πρέπει να κάνει αυτό που τις ε, επιβάλλουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι, δηλαδή η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξέρω υπάρχει κάποια παράλληλη εξέλιξη. Με άλλα λόγια, εσείς από πού παίρνετε τις ε, εντολές ε, για να εργαστείτε, για να τι εκτελέσετε. Εγώ σας είπα, πίστευα ότι παίρνετε κάποιε εντολέ και εσείς τις ε, εκτελείτε. Ε, ε, ισχύει το αντίθετο, δηλαδή εσείς έχετε μία πληθώρα ιδεών ε, και τις υποβάλλετε στους πολιτικούς για να σας πούν να τι εκτελέσετε. Και τελευταία παρατήρησή μου που αφορά στα οικονομικά. Εδώ στην Υποεπίτροπη συζητάμε βέβαια για το ότι σε σχέση με τους ε, ανταγωνιστές μας, εμείς εδώ ε, σε όλα αυτά που γίνονται τους δίνουμε την ε, μη στρατιωτική χρειά. Μετά βέβαια πολλές φορές εκπλησόμεθα όταν μπαίνουμε στο χρηματοδοτικό γιατί οι ανταγωνιστές μας από την αρχή έχουν ξεκινήσει με στρατιωτική προσέγγιση. Και όσον αφορά το μη στρατιωτικό στοιχείο αυτό ήταν ε, μια, ε, ένα παράπλευρο όφελος, έτσι θα το χαρακτηρίσω. Άρα βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση. Εσείς λοιπόν πιστεύετε ότι η πολιτική βούληση που υπάρχει μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστούν αυτές οι δύο διαφορετικές πλευρές, η στρατιωτική με τη μη στρατιωτική, στην πράξη. Πολύ εύστοχη ερώτηση, Μιχαήλ. Μην ξεχνάτε ότι 80% των εκτοξευτών, των ευρωπαϊκών εκτοξευτών, είναι εμπορική και μη στρατιωτική φύση. Το αντίστροφο συμβαίνει στι Ηνωμένε Πολιτείε, που οι περισσότεροι εκτοξευτέ μάλλον είναι στρατιωτικοί. Ο κύριο Γουαλτιέρη. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ τους τρεις ομιλητές ε, για τις ε, τόσο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους και με πυκνές ενδείξεις και προσανατολισμούς πολιτικούς. Όπως υπόθηκε κατά την πρώτη παρέμβαση, το πλαίσιο της, που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας αναδεικνύει κάποιες ασυμμετρίες στον σημερινό θεσμικό μηχανισμό, στην αρχιτεκτονική της ε, διαστημικής πολιτικής και των εμπλεκόμενων πλευρών. Έχουμε το Συμβούλιο για το Διάστημα, υπάρχει όμως και το Συμβούλιο, ο νέος η νέα αυτή μορφή του Συμβουλίου που θα ασχολείται με το διάστημα. Μετά υπάρχει το Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων Έπειτα έχουμε το διακυβερνητικό Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος που λειτουργεί επί τη βάση της ομοφωνίας. Ωστόσο ο πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται μένα από το Συμβούλιο αλλά είναι ένα, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει έτσι ένα περίεργο θεσμικό πλέγμα, μάλλον ένα πολλαπλό θεσμικό ε, πλέγμα με πολλές ισορροπίες. Και πρέπει λίγο να δούμε, να μας πείτε ίσως αυτό το θεσμικό πλέγμα πώς θα οργανώσει αυτόν τον θεσμικό αστερισμό και στο πλαίσιο της συμφωνίας πλαίσιο. Έπειτα ακολουθεί ένα ζήτημα το οποίο αφορά την βεβαιότητα των πόρων. Αναμφίβολα είναι προγράμματα βαριά, σκέφτομαι ιδίω τον Καλλιλέο, ε, ζωτικής φύσεως από πολιτική άποψη και από άποψη ασφάλειας, κοινοτικά λοιπόν προγράμματα μεγάλης σημασίας, αλλά Νομίζω ότι σε αντίθεση με άλλα προγράμματα υπάρχει μια αβεβαιότητα για το χρηματοδοτικό πλαίσιο. Πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την κατάσταση. Ε, κατά τη γνώμη σας ε, ε, είναι κάτι που πρέπει να προκαλέσει ανησυχίες ή όχι. Όπως ξέρετε το Κοινοβούλιο αγαπά πολύ το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Έπειτα υπάρχει αυτό το ζήτημα των, ε, της σχέσης μεταξύ του προγράμματος Μωυσής και του GMS. Και πάλι θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα από τεχνική άποψη. Ασφαλώς, ε, συγγνώμη όχι το Μωυσής, το Μούζης, το πρόγραμμα Μούζης. Ε, από την άλλη πλευρά πρέπει να μας ανησυχήσει λίγο η απουσία διατάξεων, προβλέψεων για τις συνεργίες που πρέπει να υπάρχουν για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την αμοιβαία οικοδόμηση σωστών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ όλων των προγραμμάτων που υπόκεινται στο ΜΟΥΖΙΣ και του GMS να καλυφθούν όλες οι όψεις και οι στρατιωτικοί. Από τεχνική άποψη ποια είναι τα προβλήματα και από πολιτική άποψη ποια είναι τα προβλήματα. Και τελευταία ερώτηση για το ζήτημα της ε, αυξανόμενης τάσης για εξωτερικοποίηση των, ή ιδιωτικοποίηση των ε, δορυφορικών συστημάτων. Ε, ακόμα και στον τομέα της ασφάλειας. Υπάρχει από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών ε, η ανάγκη για τις... Ε, ε, πώς, πώς θα διαχειριστούμε όλα αυτά τα πράγματα, τις δορυφορικές επικοινωνίες και στις σχέσεις μας με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Κυρία Γκόμες, καταρχήν θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ επίσης τους προσκεκλημένους μας για τις πολύ χρήσιμες παρουσιάσεις που μας έκαναν. Έχω τις εξής ερωτήσεις. Η χρηματοπιστωτική κρίση βλέπετε να έχει επηρεάσει και τις δικές σας δραστηριότητες και με ποιο τρόπο, με θετικό ή με αρνητικό. Θα μπορούσε ακόμη και θετικός να είναι ο αντίκτυπος γιατί ίσως τώρα αντιλαμβάνονται καλύτερα τα κράτη-μέλη την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ τους και άρα της, ε, του συνδυασμού των πόρων και τη συγκέντρωση των πόρων. Αλλά μάλλον η πρώτη αντίδραση μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση ήταν ε, αμφισβήτησης ε, των δρομολογουμένων προγραμμάτων. Ρωτώ λοιπόν, πώς ε, προχωρεί η χρηματοδότηση του προγράμματος Γαλιλαίου. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε σκληρή μάχη και είναι και διτεθειμένο στο μέλλον να συνεχίσει την προσπάθεια για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του Γαλιλαίου. Επίσης, στο ψήφισμα του Μαρτίου, επευκαιρία της έκθεσης για το διάστημα, για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προτείνει το γεωσκοπικό πρόγραμμα, το GMES, παρακολούθησης περιβάλλοντος και ασφάλειας, θα πρέπει να ασχοληθεί με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου άμυνας και ασφάλειας. Και σίγουρα από αυτή την άποψη το κέντρο δορυφόρων θα ήταν ε, ένα σημαντικός συνομιλητής στο θέμα αυτό. Επίσης, αναφέρθηκε το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται κυρίως σε εμπορική χρήση δορυφόρων και εικόνων. Αλλά στο ψήφισμά μας είχαμε ζητήσει περισσότερες συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για να διευκολύνουν πρόσβαση σε κυβερνητικές εικόνες Υπήρξε πρόοδο στον τομέα αυτό. Και άλλη ερώτηση. Εσείς παρακολουθείτε καθόλου τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο διάστημα. Η... Το Συμβούλιο σας έχει ζητήσει τη γνώμη σας ή έχετε διαμορφώσει εσείς γνώμη για αυτό το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας που προτείνεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Είναι από τεχνικά άποψη και θα καλύπτει αυτό το σύστημα αντιπυραυλικής προστασίας ολόκληρη την Ευρώπη, όλη την υπηρετική Ευρώπη ή μόνο τις χώρες του ΝΑΤΟ. Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Διαστήματος. έχει περάσει ποτέ καθόλου, κυρία Άστον, έχει παρακολουθήσει ποτέ τις εργασίες αυτού του Συμβουλίου Διαστήματος. Είχε την ευκαιρία μέχρι τώρα να το κάνει. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ναζά πρώτα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω καταρχήν φυσικά. Το Συμβούλιο Διαστήματος ίσως ε, δημιουργήθηκε κάποια σύγχυση, γιατί έχουμε δύο διαφορετικά Συμβούλια Διαστήματος. Έχουμε καταρχήν το Ιστορικό Συμβούλιο Διαστήματος, διαστήματος που προκύπτει τη Συμφωνία Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος δηλαδή είναι το Συμβούλιο του ΕΖΑ σε υπουργικό επίπεδο και το Συμβούλιο της Ένωσης από, την πλευρά της Ένωσης είναι το Συμβούλιο Ανταγωνισμού από την πλευρά του ΕΟΔ είναι οι υπουργοί που είναι αρμόδιοι για θέματα έρευνα, έρευνα διαστήματο, αλλά μπορεί να είναι και υπουργοί βιομηχανία ή οικονομία για ορισμένε χώρε. Γενικώ είναι υπουργοί έρευνα, αλλά όχι πάντα, όχι για όλε τι χώρε μέλη. Οπότε, αυτό το κοινό συμβούλιο, το μεικτό συμβούλιο διαστήματο, ε, απαρτίζεται από υπουργού 29 χωρών, δηλαδή των 27 χωρών μελών της Ένωσης ε, και των δύο χωρών Τη Ελβετία και τη Νορβηγία, που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματο, αλλά όχι και μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και το νέο όμω Συμβούλιο Διαστήματο, που είναι το Συμβούλιο Ανταγωνισμού που έχει προσθέσει στο σχηματισμό του στι αρμοδιότητέ του και το διάστημα. Απαρτίζεται φυσικά από 27 χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπουργοί ε, των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως είπε και η Σίλβια, είχαμε και την συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας για το διάστημα, στο, στην οποία ομάδα θα προσκληθεί και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ως παρατηρητής. Είναι δύο διαφορετικά λοιπόν τα Συμβούλια Διαστήματος. Το ένα είναι από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άλλο είναι συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματο και απαρτίζεται από 29 μέλη. Σε ό,τι αφορά τι αναδυόμενε διαστημικέ δυνάμει, δεν είναι πια αναδυόμενε, έχουν αναδυθεί ήδη και είναι πολύ ορατέ Εμείς έχουμε φυσικά τη περισσότερη συνεργασία με, την, με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και με τη Ρωσία είχαμε συνεργασία και με την Ινδία και την Κίνα είχαμε επιστημονική συνεργασία. Για παράδειγμα πραγματοποιήσαμε μια αποστολή στη Σελήνη σε συνεργασία με την Ινδία αλλά και είχαμε και επιστημονική αποστολή με με την Κίνα. Έχουμε κάποιους δεσμούς λοιπόν και με τις ε, χώρες αυτές, αλλά προς το παρόν περιορίζονται σε επιστημονικές ε, αποστολές. Γιατί δεν έχουμε μόνο συνεργασία με αυτές τις διαστημικές δυνάμεις, έχουμε και ένα είδος άμυλας ή ανταγωνισμού. Γιατί θα θέσουν στην αγορά εκτοξευτές, εκτοξευτήρες ή και δορυφόρους. Η διαφορά Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών σε διαστημικά θέματα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από τις επιδόσεις που θα έχει στην εμπορική αγορά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, οι δημόσιε δαπάνε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 10% των αντίστοιχων δαπανών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και παρόλα αυτά έχουμε καταφέρει να ε, κατακτήσουμε 40% της παγκόσμιας εμπορικής αγοράς ό,τι αφορά τους εκτοξευτήρες, τους εκτοξευτές και τους δορυφόρους. Οπότε η, η ισχύ μας εδώ εξαρτάται από τις επιδόσεις μας στις εμπορικές αγορές που μέχρι στιγμής είναι θαυμάσεις. είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Γιατί οι ευρωπαϊκές δημόσιες προμήθειες είναι πολύ χαλαρές σε σχέση με τις ε, αμερικανικές. Γιατί στην Αμερική, ακόμη και αν δεν έχει καμία επιτυχία στην εμπορική αγορά η Αμερική είναι τόσο ε, μεγάλη ζήτηση της εχώριας αγοράς που υπερκαλύπτονται οι ανάγκες. Δεν χρειάζεται να περιμένει από την εμπορική αγορά ε, η Αμερική για να επιβιώσει. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, επιτήρησης ή παρακολούθησης του διαστήματος, σίγουρα στο μέλλον θα καλύψει και άλλα θέματα, γιατί όπως είπαμε αυτό το, το πρόγραμμα θα στηριχθεί μακροπρόθεσμα και στις εθνικές υποδομές και πολύ συχνά σε χερσαίες υποδομές όπως το γκράφ το γαλλικό ή το τύρα το γερμανικό. Και είναι μέσα αυτά τα επίγεια μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλες εφαρμογές. Πάντως εμείς στην παρακολούθηση του διαστήματος δεν καλύπτουμε τέτοιου είδους θέματα. Βέβαια, στο μέλλον τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να μας αναθέσουν και άλλες αρμοδιότητες, κάτι που δεν ισχύει προς το παρόν. Τώρα, για τη διακυβέρνηση και τον τρόπο διοργάνωσης αυτού του αστερισμού εντό εισαγωγικών, που απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διακυβερνητικές οργανώσεις, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Φυσικά είναι μεγάλη πρόκληση η συνεργασία σε τέτοιο επίπεδο και έχουμε στην Ευρώπη, και είναι και ο, αυτός είναι και ο πλούτος της Ευρώπης, ότι έχει διάφορους σχηματισμούς, αλλά δεν είναι εύκολη πάντα η συνεργασία. Έχουμε και την ε, συμφωνία πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Θα αξιολογήσουμε αυτή την έκθεση και θα δούμε αν χρειάζεται περαιτέρω αλλαγής και προσαρμογής στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την ε, Λισαβόνα. Και αυτά θα τα εξετάσουμε στα πλαίσια του 2011 και τότε θα κρίνουμε από το Μάιο του 2011 αν θα παραταθεί αυτόματα για άλλη μια τετραετία η συμφωνία αυτή πλαίσιο ή θα αναθεωρηθεί ανάλογα με, το, με την πορεία που θα έχει η, επεξεργασία, η ανάλυση αυτή τη συνθήκη. Ό,τι αφορά την εξωτερική ανάθεση δεν έχω να προσθέσω τίποτα και για τη χρηματοδότηση θα είστε μια γενική ερώτηση για τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης Μέχρι στιγμής οι συνέπειες δεν ήταν ιδιαίτερα αρνητικές, γιατί σε καιρούς χρηματοπιστωτικής κρίσης οι επενδύσεις στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και στις πολύ εξειδικευμένες θέσεις απασχόλησης είναι μια σίγουρη και αποδοτική επένδυση, γιατί έτσι θα διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και οι επιδόσεις της βιομηχανίας. Δεν έχουμε αισθανθεί ακόμη αρνητικά αυτή την κρίση. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και την ε, νιώθουμε κι εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εμπλακεί σε περίπλοκες διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών. Εμείς το 2012 θα έχουμε το Υπουργικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος όπου θα κληθούμε να αποφασίσουμε για τα νέα προγράμματα σε ένα πιο αντίξω χρηματοοικονομικό περιβάλλον και πολύ φοβάμαι ότι θα αισθανθούμε πολύ πιο έντονα τι αρνητικέ συνέπειε τη χρηματοπιστωτική κρίση. Ό,τι αφορά την ασφάλεια σε σχέση με το γεωσκοπικό πρόγραμμα παρακολούθηση περιβάλλοντο και ασφάλεια, το GMS e αναφέρθηκε και ένα πρόγραμμα, ε, μια ομάδα εργασία για τη συνεργασία στρατιωτικού και μη στρατιωτικού κλάδου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη και η πτυχή ασφάλεια, η, η ασφάλεια του GMES. Βέβαια, το GMS ε, ισχύει τώρα, το MUSIS θα είναι για αργότερα. Αλλά υπάρχουν κάποιες ε, δυνατότητες συνέργειες. Ε, θα σας τις αναφέρει ως πιο διεξοδικά ο Ροντόλφ. Αυτά και σταματώ εγώ εδώ για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα ήθελα και εγώ να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που ετέθεσαν αφορούν ε, στον προϋπολογισμό, στις επιπτώσεις οικονομικές. Και εγώ στην ομιλία μου ανέφερα ότι από τη στιγμή που ορίζουμε τις ε, προτεραιότητές μας και από τη στιγμή που υπάρχουν οι προτεραιότητες της ε, Κομισιόν προφανώς είναι σαφές ότι συστήματα όπως το Galileo και το GMS πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτού. Βεβαίως συνεχίζονται οι συζητήσεις ε, για επιπρόσθετες ανάγκες ε, χρηματοδότησης του προγράμματος Καλαίο ε, στο πλαίσιο που έχει καθοριστεί σήμερα. Εγώ δεν είμαι αρμόδια για το πρόγραμμα Γκαλιλαίο, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί υπάρχει το φόβος να σας ε, παραπλανήσω για θέματα ε, που δεν είναι επίκαιρα, δεν είναι η τελευταία εκδοχή των εξελίξεων. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται εξελίξεις για το πρόγραμμα Γκαλιλαίο. Αυτό που ενδιαφέρει είναι μακροπρόθεσμα να διασφαλίσουμε τα προγράμματα. Και επίσης ε, γίνονται και συζητήσεις ε, για το πρόγραμμα GMES, ε, το πρόγραμμα Παγκόσμιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας. Οι συζητήσεις λοιπόν αυτή τη στιγμή γίνονται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Δορυφορικό Οργανισμό και προσπαθεί να διαπιστωθεί κατά πόσον κάτω από το πρίσμα της αποτελεσματικότερης διαχείρισης από πλευράς κόστους μπορεί μπορούμε να αναζητήσουμε νέες δυνατότητες για να ε, προκύψουν επιπρόσθετα ε, κονδύλια στο πλαίσιο της ε, τρέχουσας δημοσιονομικής προοπτικής. Πάντως αυτές είναι συζητήσεις που σας λέω χρήζουν μιας πιο εντελεχούς συζήτησης και εγώ ούτε και το πρόγραμμα Παγκόσμιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος εκπροσωπώ ούτε και εκεί θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Βεβαίως ο πρωταρχικός μας στόχος όταν είπα ότι επιθυμούμε να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία ε, για την επόμενη δημοσιονομική προοπτική τα χρηματοοικονομικά που θα μας επιτρέψουν να υπάρχει μια σταθερή μακροχρόνια βάση για τα προγράμματα πράγματι η ε, προτεραιότητες που θα καθοριστούν για την επόμενη χρονιά σίγουρα θα αφορούν τα προγράμματα GMS και το πρόγραμμα Galileo αλλά όπως σας είπα και για άλλες μελλοντικές δραστηριότητες ε, και μιλάμε δηλαδή για ένα χρονικό διάστημα από τώρα μέχρι τα επόμενα 10 χρόνια θέλουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας προσφέρει τα απαραίτητα κονδύλια για να μπορούμε να στηρίξουμε καλύτερα τη χρήση διαστημικών προγραμμάτων για λόγους ασφάλειας. Βεβαίως και μας ενδιαφέρει, ενδιαφέρει να εξασφαλίσουμε τα συστήματα αυτά, αλλά μας ενδιαφέρει επίσης να προάγουμε ε, συνεργασίες και να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα διαστημικά συστήματα μπορούν πράγματι να ε, καλύψουν ε, τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής, κυρίως κάτω από το πρίσμα της ασφάλειας. Και έτσι λοιπόν φτάνω στο ερώτημα που ετέθη σχετικά με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας. Όντι, το όντι, το ανέφερα αυτό. Επιθυμούμε το πρόγραμμα της Παγκόσμιας Παρακολούθησης του το GMS, να ασχοληθεί με θέματα ασφάλειας. Ε, ξεκινήσαμε λοιπόν να προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις ανάγκες, να δούμε τι υποτίθεται ότι θα καλύψει το πρόγραμμα GMS. Πρέπει οι αποφάσεις που θα λεφτούν στο μέλλον να έχουν ξεκάθαρα κατά νου το τι ακριβώς συζητάμε ε, ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει διάλογος τόσο ανάμεσα στα κρατημέλη όσο και με άλλες, ε, ε, άλλους ευρω, άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, να συζητήσουμε μαζί τους, ε, να διαπιστώσουμε πού ακριβώς είναι απαραίτητο να εξασθεί το θέμα του διαστήματος. Τι μπορεί να καλύψει το πρόγραμμα GMS. E Είδαμε, λέχθη αυτό, ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από τη μη στρατιωτική πλευρά με μονομερή χρηματοδότηση και τι μπορούμε να κάνουμε αν ε, μπορούμε να καλύψουμε και στρατιωτικούς σκοπούς. Το κόστος θα είναι τεράστιο, ίσως αυτό να μην αρέσει στους ε, υπουργού οικονομικών, αλλά υπάρχουν και άλλες δυνατότητες αναζήτησης ε, συνεργασιών, όπως το τομέα SSA, όπου εκεί βλέπουμε ότι είναι απαραίτητο να παρέμβει και η μη στρατιωτική πλευρά. γιατί υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλη επικάλυψη των συμφερόντων της μη στρατιωτικής ε, και της ε, στρατιωτικής πλευράς. Και εφόσον μιλάμε για κάτι ε, το οποίο έχει πληγεί εξίσου από την κρίση τόσο η στρατιωτική όσο και η μη στρατιωτική πλευρά, κατά την άποψή μας πέρα από τα αρνητικά αποτελέσματα υπάρχουν και θετικά. Ότι πλέον κανείς σκέφτεται με καινοτόμους τρόπους το πώς μπορεί να παρακάμψει τους, ε, τα διοικητικά ε, εμπόδια. Βεβαίως και υπάρχουν πολιτικά κριτήρια, αλλά το θετικό της κρίσης είναι ότι τώρα πλέον υπάρχει η βούληση να αναθεωρηθούν πολλά πράγματα με καινοτόμο τρόπο, να συνδυαστούν οι προσπάθειες έτσι ώστε να προκύψουν υπηρεσίες, ας πούμε σε στρατιωτικό επίπεδο ε, παροχή υπηρεσιών σε είδος ε, συνεργασία ε, με φορείς ε, από το στρατιωτικό τομέα που θα μας βοηθήσουν να συνδυάσουμε συστήματα ε, με φορείς από το μη στρατιωτικό τομέα. Εδώ θα σταματήσω. Παρακαλώ. Ορισμένες από τις απαντήσεις καλύφθηκαν είδος από τις συναδέλφους εδώ. Ε, οι ερωτήσεις ήταν πολλές. Θα προσπαθήσω απλώς να συμπληρώσω την εικόνα με κάποιες ε, πτυχές που είναι πολύ ευαίσθητες, όπως αφορά την πυραυλική άμυνα, ζήτημα που αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο και από τον Αντιπρόσωπο της Ισπανίας τον Ιταλό αντιπρόσωπο, συγγνώμη, τον αντιπρόσωπο της Ιταλίας. Η πυραυλική άμυνα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, όχι τόσο στη δική μας ατζέντα, όσο στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Και γιατί, γιατί εμείς στο πλαίσιο της διακυβέρνησης ανα, υπαγόμαστε, μάλλον αναφερόμαστε στα Υπουργεία Άμυνας και δεν έχει δοθεί καμιά εντολή σε εμά να έχουμε τέτοιες δραστηριότητες. Εξακολουθεί να ανήκει λοιπόν στην αρμοδιότητα των ε, κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη μπορούν να παραπέμψουν ή να αναθέσουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας τέτοια πράγματα. Ελάχιστα ε, ευρωπαϊκά κράτη θέλουν να ανοιχτούν σε κάποια ομάδα συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. αυτό είναι πολύ σαφές αυτή τη στιγμή, αλλά σας ευχαριστούμε που θίξατε το θέμα. Όσο αφορά τώρα την παρατήρηση της γης, ερχόμαστε στο ζήτημα του, της Ιταλίας και της ε, Ισπανίας, ε, τη ε, συνεργασία μεταξύ του GMES και του MUSIS. Ξεκινήσαμε από εντελώς ξεχωριστή βάση. δύο προγράμματα τα οποία έχουν διαφορετική προθεσμία, διαφορετικό χρονοδιάγραμμα και διαφορετικό διαφορετική ατζέντα. Από ό,τι καταλαβαίνω, νομίζω το γεγονός ότι δεν ξεκίνησαν από κοινή βάση ε, καθιστά δύσκολη την αναζήτηση συνεργειών. Ε, τις αναζητούμε αυτές τις συνέργειες, αλλά είναι περιορισμένης εμβέλειας. Επίσης έχουμε αντλήσει μαθήματα για τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον. Λόγω, ε, γιατί ο κύκλος των προγραμμάτων παρατήρησης της γης είναι πολύ σύντομος, γιατί οι δορυφόροι δεν έχουν διάρκεια ζωής πάνω από 4-5 χρόνια και η συζήτηση... Ε, εξακολουθεί να είναι επίκαιρη για τους επόμενους δορυφόρους. Το GMES καλύπτει πάνω από μια δεκαετία και μετά το Μούζης θα αλλάξει το τοπίο. Θα, θα υπάρξουν καινούργιοι δορυφόροι και θα χρειαστούν καινούργια οικονομικά στοιχεία, καινούργιοι μηχανισμοί. Αν δεν μπορέσουμε από τώρα να διακρίνουμε ποιες θα είναι οι συνέχειες ε, βραχυπρόθεσμα, αυτό θα κρίνει την επιτυχία των επόμενων γενεών δορυφόρων και μέσων. Όσο αφορά την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες, ε, δεν θυμάμαι αν η ερώτηση προήλθε από την Ισπανία ή την Ιταλία, η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες ε, είναι σίγουρα μια σαφή στάση στις δορυφορικές επικοινωνίες καθώς και στα παρατηρητήρια της γης. Αυτό που έχει σημασία είναι η διακυβέρνηση, δηλαδή πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχει την πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους. Και είναι πράγματι ζήτημα μεγέθους της αγοράς όσο πιο πολλά μπορούμε να, όσο περισσότερους χρηματικούς μπόρους διαθέσουμε, τόσο καλύτερο έλεγχο μπορούμε να έχουμε. Και τη στρατηγική αυτή ακολουθούν ήδη οι Ηνωμένε Πολιτείε. Η Ευρώπη πάλι ακόμη δεν την έχει ολοκληρώσει την ε, στρατηγική αυτή, γιατί η αγοραστική δύναμη της μιας κυβέρνησης είναι πολύ χαμηλότερη στην Ευρώπη από ό,τι στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και η Ζεραλντίν το τόνισε αυτό τόνισε η προσπάθεια χρειάζεται από την πλευρά των κυβερνήσεων για την στήριξη της διαστημικής πολιτικής στους τομείς της παρατήρησης της γης των δορυφορικών επικοινωνιών. Μπορούμε να λέμε ότι παίζουμε έναν ρόλο, αλλά πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι και από την πλευρά της ζήτηση. Η ανάθεση σε τρίτους συνεργάτες, εξωτερικούς συνεργάτες, μπορεί να είναι καλό ή κακό. Μάλλον δεν είναι καλό ή κακό, είναι ένα απλώς ένας τρόπος λειτουργίας. Αυτό που έχει σημασία είναι τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εγγυημένους πόρους, να διατηρήσουν κάποιο είδος ε, λαϊκής κυριαρχίας, αλλά και κάποια εγγύηση πρόσβασης. Ε, σίγουρα αυτό είναι μια τάση ε, σε επιχειρήσεις και λειτουργίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς ε, όλο και περισσότερο. Τώρα, για τις άλλους τύπους συνεργασίας, λέμε ναι σε αυτούς, γιατί θέλουμε μεγαλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γι' αυτό είμαστε εδώ, να το προάγουμε αυτό, να προάγουμε κάποιες τέτοιες ιδέες να δημιουργήσουμε και κίνητρα ε, προς μια ομάδα κρατών μελών να συνεργαστούν και από την άλλη πλευρά ε, βλέπουμε και την έκφραση του προστατευτισμού. Με συγχωρείτε. Τα εθνικά συμφέροντα ανακύπτουν στην εθνική νοοτροπία και το διαμήρασμα των ε, πληροφοριών ίσως είναι πολύ ευαίσθητο στοιχείο για κάποιες χώρες που έχουν μακρά διαδρομή εθνικών διαστημικών πολιτικών. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο αφορά τη διαστημική πολιτική δεν έχει πίσω της μακρά ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν. Και πάλι το ζήτημα έρχεται στο θέμα της διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής ε, αμυντικής ε, βιομηχανίας. Και αυτό έρχεται στο ερώτημα που μας έθεσε η Γερμανία. Ναι, έχουμε την ειδική διακυβέρνηση και εργαζόμαστε πάνω σε θέματα εθνικών υπουργείων. Μάλλον εργαζόμαστε πάνω στα θέματα για τα οποία μας δίνουν εντολή τα εθνικά υπουργεία άμυνας. Ε, εμείς προτείνουμε κάποιες ιδέες επίσης. Είμαστε δεξαμενοί σκέψεις κατά κάποιον τρόπο. Οι ιδέες αυτές πρέπει μετά να τύχουν να επενδυθούν με ισχυρή πολιτική βούληση, πράγμα που δεν το βλέπουμε ακόμα στον τομέα του διαστήματος. Δεν ισχύει ακόμα εκεί. Merci. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ε, θέλω να λάβουν το λόγο άλλοι συνάδελφοι σε σχέση με τις απαντήσεις που δόθηκαν. Ωραία. Αφού δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, ολοκληρώνουμε τη συζήτηση. Ευχαριστούμε τους προσκεκλημένους. Ήταν πολύ χρήσιμες αυτές οι παρεμβάσεις. Μην ξεχνάτε την ε, συνδιάσκεψη που γίνεται σήμερα και αύριο στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα το διάστημα. Και θα ήθελα να παροτρύνω όσους ήταν παρόντες σήμερα και συμμετείχαν στη συζήτηση να μεταβούν και αύριο στη δεύτερη μέρα της συνδιάσκεψης. Είναι αρκετά περίπλοκη η μέρη σε διάταξη γιατί και η Επιτροπή Εξωτερικών έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αύριο συνεδρίαση αλλά και τα θέματα ασφάλειας και άμυνας της διαστημική πολιτική είναι ενδιαφέροντα κάτι που θα εξετάσει η αυριανή συνδιάσκεψη, όπως σας είπα. Σας ευχαριστώ πάντως για την παρουσίαση. Το δεύτερο σημείο της σας διάταξης προβλέπει τη συζήτηση έκθεσης ΕΛΕΡ για την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία. Αυτή τη στιγμή βέβαια είναι σε μια ψηφοφορία στην Επιτροπή Ήτρε, ο Κριστιαν. Θα έρθει σε λίγα λεπτά, γι' αυτό σας προτείνω στο μεταξύ να ασχοληθούμε με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά την ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής πολιτικής. Η κυρία Ναγκόμες είναι η εισηγήτρια της έκθεσης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών που είναι επί της ουσίας αρμόδια. Εμείς ε, με την κυρία Λέζινγκ θα υποβάλουμε μια γνωμοδότηση. Στις 13 Σεπτεμβρίου μας έχει υποβάλει το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρία Λέζινγκ. Έχουν κατατεθεί 49 τροπολογίες στο σχέδιο αυτό και έγιναν ήδη εκτενείς συζητήσεις. Αν δεν έχετε αντίρρηση θα πρότεινα τώρα να εξετάσουμε την γνωμοδότηση της κυρίας Λέζινγκ. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι όσοι έχουν καταθέσει τροπολογίες, ε, κανείς από αυτούς δεν είναι εδώ. Και πριν από λίγο ε, επικοινώνησα με την εισηγητρία. Τώρα τους πράσινους ε, αυτό τους θίγει και θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ λυπηρό. Θα ήθελα λοιπόν... να πω την άποψή μου και οι ενδιαφερόμενοι να την ακούσουν. Θα εξηγήσω και πώς σκοπεύω να συμπεριφερθώ. Έτσι τώρα το να τα πω τώρα χωρίς να υπάρχει κανείς από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τι νόημα έχει. Δεν έχει νόημα. Αντιλαμβάνομαι τον προβληματισμό σας, αλλά έχουμε εδώ εκπροσώπους όλων των πολιτικών ομάδων. Και αν ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί εδώ είναι ακριβώς για να μεταφέρουν στους συναδέλφους τους ε, τα όσα θα συζητήσουμε. Και έχουμε και τους συνεργάτες, υπάρχουν βοηθοί στην αίθουσα. Οπότε δεν θα πέσει το κενό τα σχόλιά σας. Θα ληφθούν υπόψη από τις πολιτικές ομάδες, η κάθε μία θα οργανωθεί όπως το κρίνει απαραίτητο και θα διαβιβάσει περαιτέρω τις ε, απόψεις σας στους ενδιαφερόμενους. Εγώ θα έλεγα, κύριε Λέζινγκ, να μας παρουσιάσετε τη γνώμη σας για τις τροπολογίες και γύρω σε 11, 11 και 4 υπολογίζω ότι θα έρθει και ο κύριος Σέλερ μόλις ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στην Επιτροπή Ήτρε. Θα πρότεινα λοιπόν κυρία Λέζινγκ να συζητήσουμε τη γνωμοδότησή σας. Ούτως ή άλλως ε, οι ενδιαφερόμενες πολιτικές ομάδες έχουν εκπροσώπους τους, οπότε θα διαβιβαστούν τα σχόλιά σας, μην ανησυχείτε. Εντάξει? Οπότε θα ακούσουμε πρώτα την συντάκτρια της γνωμοδότησης, την κυρία Λέζινγκ, και να μας κάνει την παρουσίαση. Και ανάλογα με τις αντιδράσεις ε, μπορεί να χρειαστεί να επανέλθουμε. Άκουσα ότι ο κύριος Πιτικόφ ε, σήμερα έτσι κι αλλιώς ε, δεν θα είναι στο Κοινοβούλιο. Ε, έτσι μόλις τώρα το μαθαφώ, το μαθα αυτό, κατόπιν του, θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή την εξέλιξη. Διάβασα λοιπόν πολύ προσεκτικά τις ε, τροπολογίες, πολλές εξ αυτών μπορώ να τις δεχτώ, αλλά και άλλες ε, θα τις ε, απορρίψω. Οι τροπολογίες που στηρίζω είναι συμπληρωματικής φύσεως και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό όπως αναφέρθηκε και στην πρώτη συζήτηση δεν υπήρξε κείμενο αναφοράς ε, από την ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Αναφέρομαι κυρίως στις ε, τροπολογίες 4, 27, 36 και 39 του κυρίου Παλέκης. Οι τροπολογίε 6, 14, 19 και 38 του κυρίου Πιτικόφερ. Σε αυτές αναφέρομαι. Οι 20 και 43 της κυρία Μουνιστερικής. η τροπολογία 10 και 42 του κυρίου, της κυρίας Γετεμέκη και η 35 του κ. Φαν Όρντεν. Όσον αφορά τώρα στις ε, τροπολογίες 8 για το 2 του κ. Πίτι Κόφερ, θα ήθελα να πω ότι προφανώς εμείς δεν είμαστε κατά του περιεχομένου της ε, τροπολογίας κατά την άποψή μου η διάδοση είναι κινδυνός για όλες τις ε, αναφερόμενες ουσίες και για, τους, ε, για τις χημικές όσο και για τις βιολογικές ουσίες. Γι' αυτό λοιπόν εγώ απορρίπτω αυτή την τροπολογία διότι εδώ γίνεται λόγος μόνο για πυρηνικές ουσίες και πυρηνικά όπλα. Όσον αφορά την την 26 και την 40, τις τροπολογίες αυτές, εκεί θα δηλώσω αποχή για τους εξής λόγους. Όσον αφορά την τροπολογία 5 της κυρίας Σουγή, Εκεί γίνεται λόγος για ε, διασφάλιση της μεταφοράς ε, και της αποθήκευσης ε, των ουσιών αυτών. Βεβαίως και είναι σημαντικό αυτό, επειδή όμως εμείς ως πολιτική ομάδα επιθυμούμε πλήρη αφοπλισμό, κυρίως όσον αφορά στις πυρηνικές ουσίες και τις επικίνδυνες χημικές, αυτές οι ουσίες ούτε να μεταφέρονται ούτε να αποθηκεύονται. Γι' αυτό στην περίπτωση αυτή αποχή. Όσον αφορά στην τροπολογία 26 επίσης της κυρίας Σουγή. Εγώ δεν πιστεύω ότι μη κρατικοί οργανισμοί πρέπει μόνο αυτοί να προβάλλονται. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτιμώ αυτό που λέει ο κύριος Παλέκης, ο οποίος ε, έχει το ίδιο αυτό το περιεχόμενο ε, της τροπολογίας και το παρουσιάζει ως ένα νέο σημείο. Έτσι λοιπόν οι κρατικοί παράγοντες ε, αναφέρονται σε σχέση με τη σύμβαση και σχετίζονται με αυτή. Το ότι η σύμβαση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη ε, τον κίνδυνο από μη κρατικού φορεί. Αυτό με οδηγεί στο να δηλώσω αποχή στην τροπολογία Σουγή και να δεχθώ την τροπολογία του κυρίου Παλέκης ε, που εκτός από αυτό το ένα θέμα ταυτίζονται. Η τρίτη αποχή εκ μέρου μου αφορά το εργαλείο για σταθερότητα ή την αναφορά του εργαλείου αυτού. Γνωρίζω πολύ καλά ότι όσον αφορά στο εργαλείο για τη σταθερότητα ε, μπορούν να χρηματοδοτηθούν πάρα πολλά σημαντικά πράγματα όπως ε, τα ε, μέτρα CBNR. Παρ' όλα αυτά η πολιτική μου ομάδα επικρίνει την έλλειψη διαφάνειας και απορρίπτει τη χρηματοδότηση για αυτό το εργαλείο δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ αυτής της τροπολογίας. Όσον αφορά στις υπόλοιπες τροπολογίες, αυτές είτε έχουν ως στόχο ε, το στρατιωτικό στοιχείο στην προστασία καταστροφών είτε στρέφονται κατά της εγκατάστασης μιας ζώνης ελεύθερης από πυρηνικά. Κατά την άποψή μου υπάρχουν σημαντικά αιτήματα ε, για τη μη διάδοση που διαγράφονται. Ε, κατόπιν τούτου δεν μπορώ επουδενή να στηρίξω αυτή την τροπολογία και αν αυτές οι τροπολογίες κατατεθούν θα ζητήσω το όνομά μου ε, να αφαιρεθεί από αυτές τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστώ. Θέλει κανεί το λόγο από του κοιόδης ηγητέ, η κυρία Σουλή. Ε, euh, Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή την κυρία Λέζινγκ. Είναι σαφές ότι η γνωμοδότησή της έχει μια έντονη πολιτική χαριά. Αλλά δεν είναι και πολύ ρεαλιστική αυτή η γνωμοδότηση, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τον ε, ακριβή στόχο. Δηλαδή να βοηθήσει τον πληθυσμό σε περίπτωση ατυχήματος ή απόπειρας CBRN. Το θέμα της μεταφοράς και της αποθήκευσης, όπως είπε η κυρία Λέζινγκ, είναι κέριο. Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές ασφάλειας για τη μεταφορά και την αποθήκευση. Έτσι θα έχουμε λιγότερους κινδύνους ε, ε, υπεξαίρεση τέτοιου υλικού. Επίσης, ε, Είχαμε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί και σε ό,τι αφορά τα... την έκκληση για τον πυρηνικό αφοπλισμό δεν νομίζω ότι έχει θέση σε αυτή τη γνωμοδότηση. Σε ό,τι αφορά την διαπεριφερειακή συνεργασία νομίζω είναι ένα πολύ κατάλληλο επίπεδο για τη συζήτηση αυτή και τονίσαμε και την ανάγκη ενίσχυσης της στρατητικη συνεργασίας. Είναι αδύνατον να είμαστε αποδοτικοί και αποτελεσματικοί αν στερηθούμε αυτή τη συνεργασία και ιδιαίτερα το στρατιωτικό κλάδο που έχει πείρα σε θέματα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά κτλ. Επίσης, ζητούμε ενίσχυση των δυνάμεων πολιτικής προστασίας και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Η έκθεση της ουσίας της κυρίας Γκόμες είναι καταπληκτική, εξισορροπημένη, λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές αυτού του ζητήματος. Κρίμα θα ήταν λοιπόν να την αλλοιώσουμε με μια γνωμοδότηση σαν αυτή τη κυρία Λέζινγκ. Σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε Μπιτικόφερ και τι δικέ μου, εγώ δεν έχω βρει διαφορέ μεταξύ του. Είμαι συγγνώμη, σε ό,τι αφορά την τροπολογία 27 του κυρίου Παλέσκης και 26 τη δικιά μου, πραγματικά πρέπει κανείς με μεγεθυντικό φακό να ψάχνει τις διαφορές. Εγώ δεν βλέπω μεγάλες, δεν βλέπω διαφορές μεταξύ των δύο τροπολογιών. Η κυρία Γκόμες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις προλαλήσεις σας, την κυρία Λέζιν και την κυρία Σουγή Ίσως το γεγονός ότι η κυρία Λέζινγκ συνέταξε την γνωμοδότησή της πριν καταθέσω εγώ το σχέδιο έκθεσής μου, ίσως ε, την περιόρισε. Γιατί όπως είπε η κυρία Σουγή, όντως ε, η έκθεσή μου είναι πολύ ευρύτερη από τη γνωμοδότηση. Και είναι πολύ ευρύτερη το θέμα του αφοπλισμού. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι μια γνωμοδότηση της Υποεπιτροπής ε, Ασφάλειας και Άμυνας ε, λαμβάνει υπόψη και το θέμα του αφοπλισμού, αλλά ο αφοπλισμός δεν είναι το επίκεντρο της έκθεσης, ούτε ο κύριος στόχος της έκθεσης. Εμείς προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους κινδύνους και τις απειλές, προσπαθούμε να προετοιμαστούμε για να τις αποτρέψουμε και επίσης εξετάζουμε το ενδεχόμενο αντίδρασης ε, προκειμένου να προστατεύσουμε τον πληθυσμό από τέτοιες απειλές. Εγώ στην έκθεσή μου ήδη έχω συμπεριλάβει κάποιες ε, ιδέες της γνωμοδότησης ε, Λέζινγκ που αφορά τον αφοπλισμό μόνο. Αλλά διαφωνώ με την προσέγγιση της ε, εισηγήτριας. Διαφωνώ με την πρόταση για αποκλεισμό της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας. Γιατί για μένα αυτή η συνεργασία είναι νευραλγικής σημασίας. Για να έχουμε ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό σύστημα αντίδρασης και αποσόβησης τέτοιων απειλών, χημικών, βιολογικών και ραδιολογικών όπλων, μια αποτελεσματική αντίδραση στηρίζεται σε αυτή την πολιτικοστρατητική συνεργασία, κατά τη γνώμη μου. Και ήδη από τον περασμένο Ιούλιο υπάρχει αυτή η πρόταση από το Συμβούλιο. Οπότε είναι κρίμα να αστερηθούμε αυτή την πολύ σημαντική διάσταση της ε, πολιτικο συνεργασίας. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της ενίσχυσης. Συμφωνώ με τις προτάσεις της κυρίας Σουγή για πολλές τροπολογίες που είναι πανομοιότητες. Παλέτσκι, Μπουτικόφερ, Σουγή, και είμαι υπέρ τη ε, ενίσχυση τη διαπεριφερειακή συνεργασία που έχει κεφαλαιώδη σημασία και επίση υπέρ τη ενίσχυση των δυνάμεων πολιτική προστασία. Στην Πορτογαλία ε, διοργανώσαμε μία δημόσια ακρόαση για την αξιολόγηση του τρόπου εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράση από τι εθνικέ αρχέ. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο αυτό, γιατί κάθε χώρα είναι ένα κρίκο αυτή τη αλυσίδα και άλλωστε έπρεπε να ξεκινήσω κι εγώ από την πατρίδα μου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι, όλες οι αρμόδιες αρχές και οι πολιτικές και οι στρατιωτικές γνώριζαν την ύπαρξη του σχεδίου δράσης, κάτι που είναι πολύ θετικό και μάλιστα μερικοί είχαν συμμετάσχει κιόλα αυτή την, στην κατάρτιση, στην εκπόνηση αυτού του σχεδίου δράσης. Αλλά το πιο σημαντικό συμπέρασμα αυτής της δημόσιας ακρόσης είναι ότι δεν υπάρχει μία κεντρική εθνική αρχή που θα εξασφαλίζει το συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Ακόμη και σε επίπεδο πληροφοριών, συγκέντρωση πληροφοριών, intelligence και διάδοσης ε, των διαβαθμισμένων πληροφοριών, των απόρριτων πληροφοριών που χρειάζονται πολλές φορές ε, οι αρχές για να αντιληφθούν ε, τους κινδύνους και τις απειλές και να ετοιμάσουν την αντίδρασή τους. Υπήρξαν βέβαια και άλλες πτυχές Μερικές φυσικά ήταν πιο εθνοκεντρικές ό,τι αφορά την προετοιμασία αυτού του σχεδίου δράσης. Πάντως ήταν πολύ ενδιαφέρον που ήδη έχουμε παρουσία σε ευρωπαϊκές, πανευρωπαϊκές ασκήσεις και η συμμετοχή αυτή είναι πολύ χρήσιμη. Υπάρχει και το θέμα της ενίσχυσης των δυνάμεων πολιτικής προστασίας, που επίσης είναι κέριο. Είμαστε αναφανδόν υπέρ αυτής της ενίσχυσης Κάτι που απαιτεί όμως μία ιδιαίτερη προετοιμασία σε περίπτωση που μιλούμε για τέτοιες ουσίες χημικές, βιολογικές, ε, ραδιολογικές ή πυρηνικές, γιατί οι ουσίες αυτές προϋποθέτουν μία κατάρτιση, μία ειδική προηγούμενη εξάσκηση και προετοιμασία. Τώρα το θέμα της ε, προσπάθειας αντιμετώπισης ή ε, αντίδρασης, τροπολογία Παλέτσκης, το επισημαίνω και εγώ στην έκθεσή μου, γιατί η χρησιμοποίηση αυτών των ουσιών δεν έχει μόνο στρατιωτικό χαρακτήρα και εργαστήρια οι τις χρησιμοποιούν και κάποια ερευνητικά κέντρα τις χρησιμοποιούν. Ακόμη και επιχειρήσεις. Γιατί ξεχνάτε ότι μιλούμε για χημικές και βιολογικές ουσίες που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά. Οπότε θα πρέπει να εφαρμόσουμε όλες τις συνθήκες που διέπουν αυτές, τη χρήση αυτών των ουσιών, ώστε να ελέγξουμε την πρόσβαση σε ουσίες αυτές ανθρώπων που θα είναι καταρχήν προσδιορισμένοι, εντοπισμένοι, μπορούμε να τους ε, ταυτοποιήσουμε και φυσικά να οριοθετήσουμε την ε, πρόσβαση σε τεχνολογία που μπορεί να παρεκτρέψει τη χρήση αυτών των ουσιών για τρομοκρατικές απειλές ή τρομοκρατικές ενέργειες. Θα πρέπει να περιορίσουμε αυτή τη χρήση, αλλά έχουμε φυσικά και άλλες θεομηνείς φυσικές καταστροφές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Είχαμε πρόσφατα την οικολογική καταστροφή στην Ουγγαρία με την ερυθρά υλή, τα τοξικά αυτά απόβλητα, την κόκκινη λάσπη και είναι χαρακτηριστική περίπτωση χημικής καταστροφής. Καταστροφής δηλαδή χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής υφής και μάλιστα δεν, δεν γνωρίζουν σύνορα τέτοιου είδους καταστροφές. Ξεπέρασαν στην περίπτωση αυτή τα ουγγρικά σύνορα και χρήζουν μίας παρέμβασης όχι μόνο εθνικής αλλά και περιφερειακής και πανευρωπαϊκής. Στην περίπτωση της Ουγγαρίας μάλιστα ήταν ενδιαφέρον γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμέσως μετά το αίτημα της Ουγγαρίας ενεργοποίησε το μηχανισμό άμεσης αντίδρασης με την στρατολόγηση εμπειρογνωμόνων, την κινητοποίηση εμπειρογνωμόνων προκειμένου να βοηθήσουν τις αγγρικές αρχές να προσδιορίσουν την έκθεση των ζημιών και να θεσπίσουν κάποια μέτρα μετριασμού τους και περιορισμού τους. Αρκετές τροπολογίες κατα... κατατέθηκαν για την ε, γνωμοδότηση Λέζινγκ. Ήδη πολλές καλύπτονται από τη δική μου έκθεση που ακολούθησε την υποβολή της γνωμοδότησης κυρίας Λέζινγκ όπως σας είπα. Και φυσικά είμαι πρόθυμη να λάβω υπόψη τις προτάσεις των συναδέλφων και φυσικά και της ίδιας συγκήτριας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να παρέμβουν άλλοι συνάδελφοι. Ο κύριος Παρέτσκης, ο οποίος έχει υποβάλει και πολλές τροπολογίες. Ε, ως προς τις τροπολογίες μου, έχω προτείνει ε, εκείνοι που προτείνουν τακτικές αξιολογήσεις κινδύνου στον τομέα των χημικών, βιολογικών, τεχνολογικών και πυρηνικών ουσιών ε, καθώς και εκείνοι που εκπονούν μέτρα ανταπόκρινσης και αντιμετώπισης και κυρίως ε, ιατρικά μέτρα και παραθέτω ε, καλούν τα κράτη-μέλη και την ε, Επιτροπή να προτείνουν βέλτιστες λύσεις και να απευθύνονται στους κατάλληλους εμπειρογνώμονες. Επίσης, τακτικές ε, αναφορές να υποβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβόλιο για την εκτίμηση και διαχείριση του χημικού, βιολογικού, κτηνολογικού και πυρηνικού κινδύνου προτείνω να διοργανωθεί μια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να, να κληθούν αντιπρόσωποι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ε, σχετικούς κλάδους αυτό δεν είναι τροπολογία, είναι μια υπόδειξη, μια πρόταση. Και γενικά θέλω να τονίσω ότι το να είμαστε προετοιμασμένοι για όλους αυτούς τους κινδύνους και τις επιθέσεις ε, είναι κάτι που ποικίλει πάρα πολύ από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και ιδίως τα καινούργια κράτη-μέλη δεν είναι τόσο καλά προετοιμασμένα για τέτοια ενδεχόμενα. Όπως ξέρουμε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η καλύτερη χώρα μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών χωρών, αλλά σε γενικές γραμμές ε, είμαστε πολύ πίσω σε σύγκριση όχι μόνο με τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά ακόμη και με μερικές ασιατικές χώρες. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα λοιπόν και η έκθεση αυτή είναι μια πολύ σημαντική έκθεση. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Έλμς. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Παρακαλώ, η κυρία Λόζη πάρα πολύ γρήγορα θα ήθελε ίσως να προσθέσει κάτι στην ε, συζήτηση. Θα θέλατε, αλλά πολύ γρήγορα, παρακαλώ. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Θα περιμένω τις συζητήσεις μέχρι το τέλος. Υπάρχουν πάρα πολλές γνώμες από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, περνάμε στην ε, έκθεση για την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία και την ανάπτυξη στρατιωτικών ε, ικανοτήτων. Είναι μια έκθεση που θα συζητηθεί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων την Πέμπτη. Υπάρχουν, ε, έχουν υποβληθεί 55 τροπολογίες. Ο κύριος Έλλερ προτείνει 11 συμβιβαστικές τροπολογίες. Ίσως μπορείτε να μας παρουσιάσετε εν συντομία που βρισκόμαστε. Πολύ γρήγορα παρακαλώ. εγκάρδιες ευχαριστίες. Ε, ζητώ συγνώμη για την ε, καθυστέρηση, αλλά στην Ήτρε ψηφίζαμε για την ε, ενεργειακή στρατηγική για το 2011 και μετά. Ζητώ λοιπόν συγνώμη για την αργοπορία μου. Περνάω στα αγγλικά. Ευχαριστώ όλες τις ομάδες. Πιστεύω ότι είχαμε μια πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και πολύ γόνιμες μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Πιστεύω λοιπόν ότι η έκθεση γενικώ προχωράει σε σωστή κατεύθυνση πιστεύω ότι υιοθετεί και θα παίζουν σημαντικό ρόλο οι απόψεις του Κοινοβουλίου. Έχουν ε, υποβληθεί πάνω από 150 τροπολογίες, πολλές από αυτές καλύπτονται από άλλες από την έκθεση, άλλες από άλλες τροπολογίες. Έχουμε λάβει και τροπολογίες για την ισότητα των φύλων και προσπαθούμε να ενοποιήσουμε το κείμενο προτείνοντας 12 συμβιβαστικές τροπολογίες και προτείνοντας ε, ε, και κάνοντας διάφορες προτάσεις που στόχο έχουν την συνοχή του κειμένου. Κάποιε τροπολογίε ίσω πρέπει να ενταχθούν σε άλλα τμήματα του κειμένου. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω του κοιόδη εισηγητέ και τα μέλη υπάρχει συμφωνία για ένα ευρύ φάσμα τροπολογιών. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλά διαρθρωμένη έκθεση, η συμβιβαστική πρόταση 2. Υπάρχει συχνά έντονη ανάγκη για μια πολιτικοστρατιωτική προσέγγιση στις κρίσεις και ε, και ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις ε, μπορεί να αρκεί μόνο η πολιτική ή μόνο η στρατιωτική προσέγγιση. Η συμβαστική συμβιβαστικη προταση 3 καλύπτει περισσότερο τους, τις μη κρατικούς φορείς, τις μη κυβερνητικές ε, οργανώσεις ε, στην πρόληψη των έναπλων συγκρούσεων. Η συμβαστική πρόταση 4 αφορά τις σχέσεις μεταξύ ε, επίσημων φορέων της πλατφόρμας για την κρίση και άλλες δομές, ιδίως όσον αφορά το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των χρηματοδοτικών μέτρων από το Εργαλείο για τη Σταθερότητα και συνδέσμους μεταξύ ε, των διαφόρων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των φορέων. Η συμβιβαστική πρόταση 5 αποδέχεται καταρχήν την ανάγκη μιας νέας δύναμης πολιτικής προστασίας, αλλά διευκρινίζει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί μια καινούργια μόνιμη δύναμη. Απλώς θα βασίζεται σε μια εθελοντική δεξαμενή εθνικών εθελοντών και σε έναν καλύτερο μηχανισμό λειτουργίας των υφιστάμενων των μηχανισμών πολιτικής προστασίας. Πρόταση 6, συμβιβασμός 6. Συμπληρώνει την ανάγκη για μια σωστή ισορροπία πολιτικού και στρατιωτικού για τη σωστή ολοκλήρωση των στρατηγικών πλάνων έτσι ώστε να μην υπάρξει σύγχυση μεταξύ του πολιτικού και στρατιωτικού ρόλου. 7 ο ρόλος της ΕΤΑ και το γεφύρωμα των δύο χωριστών διαδικασιών ανάπτυξης των πολιτικών και στρατιωτικών ικανοτήτων Συμβαστική πρόταση 9 ε, τροπολογίες για το ρόλο της ΕΤΑ. Ε, συμβαστική πρόταση 11 τονίζει την αρχή της λήψεως αποφάσεων, της αυτονομίας της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων σε σχέση με τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ ε, και με βάση περαιτέρω συζητήσεις θα ήθελα τώρα να σας να προτείνω και την συμβαστική πρόταση 12 για μια σαφή διατύπωση της παραγράφου 43 που έχει να κάνει με τη νέα στρατηγική άποψη του ΝΑΤΟ και σε σχέση με τις πολιτικές κρίσεις ε, θέλει να, ε, η πρόθεση μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα οδηγηθούμε σε περιττό επαναλήψεις στην ανάπτυξη των ε, στρατιωτικοπολιτικών ικανοτήτων. Νομίζω με όλες, όλες αυτές οι συμβιβαστικέ ε, τροπολογίες υποστηρίζουν την έκθεση. Είμαι πολύ ευγνώμων και θα ήθελα να αναδείξω το ρόλο ε, της γραμματείας. Εξαιρετική δουλειά ε, στο να βρει και να διατυπώσει τις προ... τους συμβιβασμούς και είμαι πολύ ευγνώμων που καταφέραμε να εντάξουμε νομίζω όλες τις θετικές προσεγγίσεις, όλα τα θετικά σχόλια από όλο το φάσμα των πολιτικών ομάδων που έδειξαν ενδιαφέρον για την έκθεση. Αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω ένα-δυο σημαντικά σημεία. Κάποιες τροπολογίες είχαν να κάνουν με τη χρήση στρατιωτικών μέσων στην ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Προάγεται η χρήση των ε, στρατιωτικών μέσων για την ε, ανακούφιση από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Υπήρχαν αντιρρήσεις από ορισμένους γιατί ε, προάγεται και η αυξημένη χρησιμοποίηση ενόπλων ε, ικανοτήτων για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων, αλλά όπως αναφέρεται σαφώς στην έκθεση, αυτό θα γίνεται μόνο στο πλαίσιο των διεθνών κατευθυντήριων γραμμών και συγκεκριμένα του Όσλο. Η χρήση ε, στρατιωτικών μέσων θα πρέπει πάντοτε να είναι η τελευταία λύση. Θα προάγονται κυρίως μη στρατιωτικής φύσεως μέτρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό συνδυάζοντα την πολιτική και στρατιωτική τη ικανότητα. Έτσι όμω χρειάζεται τις ένοπλες ομάδες, ε, γιατί πολλέ φορέ είναι χρήσιμε στην παροχή ανθρωπιστική βοήθεια. Για παράδειγμα, πρέπει να μπορούν οι αστυνομικέ δυνάμει να μπορούν να συνεργάζονται σωστά και στενά με τι στρατιωτικέ μονάδε και να στηρίζουν ε, τι πολιτικέ δράσει στον τομέα τη ανθρωπιστική βοήθεια και πάλι πάντοτε εναρμονισμένα με τι διεθνεί οδηγίες. Όσο αφορά το μέλλον αυτών των ομάδων, τονίζεται ότι απαιτείται κάποια οικονομική αλληλεγγύη, αλληλεγγύη αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μάχημες ομάδες, οι οποίες θα πρέπει να μετέχουν σε πιο μακροπρόθεσμες συνεργασίες Κάποιες τροπολογίες αφορούν την ισορροπία στρατιωτικού πολιτικού στη διαδικασία του σχεδιασμού. Θέλω να τονίσω ότι η έκθεση αναδεικνύει την έλλειψη πολιτικών εμπειρογνώμων, ιδίως στις, στους τομείς προτεραιότητας, όπως αστυνομία, διοίκηση, πολιτική προστασία. Χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό. Η μεγάλη πλειοψηφία των αποστολών είναι πολιτικής φύσεως, αλλά αυτό δεν δεν αντανακλάται στις ε, δομές μας. Αυτό που πρέπει να πετύχουμε στη μελλοντική στρατηγική είναι μια σωστή ισορροπία μεταξύ των, της και της στρατιωτικής ε, προσέγγισης να μην υπερισχύει καμία πλευρά, να μην επικρατεί καμία από τις δύο διαστάσεις. Όσο αφορά τη χρηματοδότηση της αμυντικής έρευνας, αυτό είναι ένα από τα πιο επίμαχα ζητήματα της έκθεσης. Η έκθεση προάγει την έβρεση συνεργειών και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα και των ειδικότερων τομέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι πολλές συνέργειες μπορούν να διερευνηθούν μεταξύ της αμυντικής, ε, στρατιωτική και ε, πολιτικής άμυνα. Ωστόσο δεν θέλω να ανοίξω το ζήτημα παράτασης του προγράμματος πλαισίου καθεαυτού για να καλυφθεί η αμυντική έρευνα. Κατά την άποψή μου ε, αυτό πρέπει να το αποφασίσει η συζήτηση για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο και δεν, αυτό το θέμα δεν ανήκει στις συμβιβαστικές προσπάθειες. Νομίζω ότι πρέπει να εμείνουμε σε ό,τι αποφασίστηκε πριν από πέντε χρόνια στο πρόγραμμα πλαίσιο. Ωστόσο, πρέπει να γίνει μια συζήτηση για την ε, αμυντική έρευνα. Εγώ το βλέπω να συνδέεται περισσότερο με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας παρά το αντίστροφο. Τέλος, είναι η πρόσβαση του ΝΑΤΟ στις καινούργιες πολιτικές μας ε, δυνατότητες. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει ε, να ότι πρέπει να αποφεύγεται η επανάληψη δομών και ενεργειών από το ΝΑΤΟ. Ε, θα πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση υπό ορισμένε προϋποθέσεις. Πρέπει να τονίσω ένα τελευταίο σημείο εδώ Είτε το θέλουμε είτε όχι, το ΝΑΤΟ σκέφτεται να συμμετέχει και αυτό στον τομέα διαχείρισης πολιτικών κρίσεων. Και το ΝΑΤΟ δυστυχώς λειτουργεί επί τη βάση της ε, υπόθεσης, ε, της υπόθεσης ότι δεν υπάρχει η αντίστοιχη ικανότητα στην πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα μεγάλο λάθος να αφήσουμε δηλαδή το ΝΑΤΟ να ξεκινήσει μόνο του στην ανάπτυξη πολιτικών ικανοτήτων, γιατί αυτό θα καταλήξει σε μεγάλη επανάληψη προσπαθειών. νομίζω ότι θα πρέπει ε, το, το σχέδιο έκθεσης λέει ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να μπορεί να βασίζεται στις ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον τομέα αυτού. Αυτό. Τώρα το πώς θα βασίζεται το ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Να δούμε και τη συνεργασία και με άλλους διεθνούς, διεθνείς φόρους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ε, νομίζω ότι αν ψηφιστεί αυτή η έκθεση θα έχουμε μια ισχυρή φωνή στο μέλλον στις σχετικές αποστολές. Σας ευχαριστούμε κύριε Έλερ. Πολύ μεστές οι παρατηρήσεις και εξαιρετική η έκθεση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτος σε ένα συνάδελφο που θα φύγει και με, με την άδεια του αντιπρόεδρου, στην κυρία Φρασίσκα. Ευχαριστώ πολύ. Αλλιώς τα είχα προγραμματίσει. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ ε, που πρέπει να φύγω. Και ευχαριστώ που μου δίνετε τώρα το λόγο που με προτάσετε. Εμεί ε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε για μια κατά την άποψή μας πολύ καλή έκθεση ε, που έθιξε πολλά και σημαντικά θέματα. Αναφερθήκατε και στο θέμα του ΝΑΤΟ που συμμεριζόμαστε 100% την άποψή σα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που στο συμβασμό υιοθετήσετε πολλέ δικέ μας απόψεις. Και επιτρέψτε μου να θίξω κάποια σημεία ε, για να είναι σαφή η θέση μας όσον αφορά τη συμβαστική πρόταση 4. Η πρόταση αυτή κατά την άποψή μας ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Ίσως ε, να σας μοιάζει έτσι πολύ σχολαστικό ε, που θέλω να επιμείνω σε κάποιες λεπτομέρειες αλλά εν πάση περιπτώσει πρόκειται για τα 250 εκατομμύρια σε τήσια βάση το εργαλείο της σταθερότητας και εμείς ε, αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε γιατί δεν γνωρίζουμε ποιος θα προγραμματίσει το περιεχόμενο αυτού του εργαλείου είδαμε τα έγγραφα και είδαμε ότι όσον αφορά την πλησία εξωτερική δράση, αυτή θα ασχολούνται κυρίω με την οικονομική διαχείριση. Όσον αφορά όμω το περιεχόμενο, ποιο θα κάνει το σχεδιασμό του περιεχομένου. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό ε, το Κοινοβούλιο να επισημαίνει στους αρμόδιους κομισιών ότι είμαστε αρμόδιοι και ίσως μπορούμε να αναλάβουμε ένα κομμάτι από την ε, ε, αρμόδια διεύθυνση επιτροπής. Ε, να πω δύο λόγια επ' αυτού και εάν τελικά η δική μας τροπολογία χρειάζεται υποστήριξη θα καλέσω και κάποιες άλλες ομάδες να τη στηρίξουν. Να πω και κάτι άλλο για την τροπολογία υπεριθμών 16 Ίσως αυτό ε, να σας μοιάζει ε, πολύ στήρο με αριθμούς, ε, αναφέρονται διάφοροι αριθμοί για τις αποστολές, τους αριθμούς των αποστολών. Νομίζω ότι μπορεί να υιοθετηθεί το δεύτερο κομμάτι που λέει υπενθυμίζει 16 από 24 αποστολές ε, έχουν μη στρατιωτική αποστολή υπάρχει κάποια έλλειψη ισορροπίας ε, ε, στο προσωπικό γιατί περισσότεροι είναι στρατιωτικοί. Τέλος της παράθεσης, αυτό που ενδιαφέρει είναι ποια ε, είναι η σύσταση αυτή τη, στιγμή των αποστολών, η μορφή της σύστασης, στρατιωτική ή μη. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι κατά την άποψή μου δεν είναι απόλυτα σαφές κατά πόσον μιλάμε για συγκρούσεις, αιστείες σύγκρουσης ή για ε, καταστροφές και αντιμετώπιση καταστροφών. Πρέπει κανείς να τα διαβάσει πολύ προσεκτικά ε, για να κατανοήσει περί τίνος ε, πρόκειται να μην τα μπερδέψει. Και εγώ δεν κατάλαβα καλά κατά πόσο μιλάμε για καταστροφή ή για σύγκρουση disaster ή κάποια άλλη μορφή σύγκρουσης. Μετά, πρόκειται για την εκπροσώπηση στις αποστολές. Μέχρι τώρα υπάρχει μια έκθεση ε, περσινή όπου αναφέρεται ότι το 37,5% του πολιτικού προσωπικού προέρχεται από τα νέα κράτη-μέλη. Καλό είναι αυτό, είναι το 1 τρίτο. Γι' αυτό λοιπόν ή μάλλον το θέμα δεν είναι να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να στείλουν ε, περισσότερους εκπροσώπους. Γι' αυτό καταθέσαμε την τροπολογία ότι τα κράτη-μέλη να ε, στείλουν περισσότερους εκπροσώπους αλλά οι περισσότεροι να είναι μη στρατιωτικοί. Το θέμα πολλές φορές είναι ότι δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό αλλά έλλειψη προσωπικού. Ίσως λοιπόν εδώ μπορούμε να καταθέσουμε μία προφορική τροπολογία μετά την πρώτη ανατελεία να αναφέρουμε καλή τα κράτη-μέλη να στείλει στις ευρωπαϊκές αποτολές ε, μη στρατιωτικό προσωπικό για να επικρατήσει ισορροπία. Ε, όπως σας λέω λοιπόν ε, πρέπει να σταλεί περισσότερο προσωπικό. Αυτή απλά είναι μία πρόταση. Κατόπιν, όπως σας είπα την έκθεση τη βρίσκω πάρα πολύ καλή. Ε, θα υποστήριζα όλα, αλλά για τη δική μας την πολιτική ομάδα υπάρχουν δύο θέματα επίμαχα. Το ένα είναι defensive research, αμυντική έρευνα. Αυτό, αυτή την τροπολογία μπορούμε να τη δεχτούμε, αλλά την 126, 131 και 133, οι τροπολογίες αυτές ε, για μας ε, δεν είναι αποδεκτές FP7 και FP8 ε, το χρηματοδοτικό αυτό πλαίσιο για μας δεν είναι το πλαίσιο όπου πρέπει να ενταχθεί η άμυνα. Γι' αυτό διαφωνούμε. Τα κονδύλια προβλέπονται για άλλους ερευνητικούς σκοπούς και δεν επιθυμούμε να ενταχθεί εκεί αυτή η έρευνα. Γι' αυτό λοιπόν ε, εμείς δεν θα συμφωνήσουμε με αυτή την τροπολογία. Ένα άλλο θέμα για τις καταστροφές και προστασία από τις καταστροφές και εκεί διαφωνούμε. Όπως σας είπα λοιπόν, ε, στο Κονγκό παραδείγματος χάρη, αν θέλουμε, εκεί μπορούμε να προστατεύσουμε το πολιτικό προσωπικό. Υπάρχει αρκετό πεδίο προστασίας. Δεν πρέπει αυτό απαραίτητα να γίνει σε περίπτωση συγκρούσεων στο Κονγκό που σας είπα έτσι μου ήρθε στο μυαλό αλλά κύριε Έιλερ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την καλή συνεργασία και νομίζω ότι η έκθεση είναι πολύ καλή Ευχαριστώ πολύ Πριν δώσουμε το λόγο στον Αντιπρόεδρο Μαυρό Κοράς. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια στο πλαίσιο της ιδιότητός μου ως Προέδρου ε, σε σχέση με τις βιβαστικές τροπολογίες και τη σχετική συζήτηση. Η ίδια συζήτηση έγινε κατά την επεξεργασία της έκθεσης ε, για την, για την πολιτική στρατηγική ε, άμυνας πέρυσι και ε, ξαφνιάστηκα από την καχυποψία που υπάρχει γύρω από ορισμένα εργαλεία όπως το CM5 δηλαδή την ε, μονάδα σχεδιασμού, ε, λόγω της, ε, του στρατιωτικού υπόβαθρου ορισμένων μέλων, ναι, πράγματι έχουν ένα στρατιωτικό υπόβαθρο, μα ακριβώς γι' αυτό είναι και πιο αξιόπιστοι ώρες-ώρες μπορούμε να πούμε και δεν πρέπει να ενεχοποιούνται γιατί, ήταν, γιατί είχαν κάποια προϊνστική εμπειρία. Ε, νομίζω ότι ε, τι να κάνουμε, κακό είναι να υπάρχει ανισορροπία, αλλά εξ ορισμού αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη πείρα. Τώρα, όσο αφορά τον καταμερισμό των δύο φύλων, δεν υπάρχει ανισορροπία στο διευθυντικό επίπεδο. Ε, ε, πολύ καχυποψία λοιπόν, πολλές καταγγελίες, πολλές αλληλοκατηγορίες, αλλά θα, θα να είμαι πολύ ακριβής. Ε, πρέπει πραγματικά όλοι σας να τηρούν τη σωστή ισορροπία σε επίπεδο φύλων, σε επίπεδο αρμοδιότητα, σε επίπεδο υπόβαθρου. Εντάξει, σωστά όλα αυτά αλλά να μην υπάρχουν προκαταλήψεις. πολύ φοβάμαι ότι τα σχόλια προέρχονται από προκαταλήψεις. Τέλος, χωρίς αναγκαστικά να επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες, θεωρώ επιζήμιο να, να μην αντλούμε από όλο το χρήσιμο έργο που έχει ήδη γίνει. Ασφαλώς να γίνει κάποια συμβιβαστική τροπολογία. Αλλά εγώ θα ήθελα να αναφέρεται η Επιτροπή 8 ε, και αυτή την άποψη τη συμμερίζονται και άλλοι μεταξύ μας. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Μαρόνι, ο οποίος... Τον κύριο Μαυρονικόλα, ο οποίος είναι ο σκιώδη εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή αφορά την πολιτικοστρατητική συνεργασία και ανάπτυξη των πολιτικοστρατητικών ικανοτήτων, ένα καινούριο θέμα δηλαδή, θα ήθελα να υπογραμμίσω την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με τον Κρίστιαν Έλερ και κάποιες επαφές στις οποίες καταφέραμε να συμπεριλάβουμε πολλές από τις τροπολογίες στην έκθεση. Μετά από τις συνεννοήσεις και επαφές που είχαμε με τον εισηγητή αποφασίσαμε να αποσύρουμε 19, 23, 34, 100, 23 και 43. Πολλές τροπολογίες συμφωνήσαμε να τις αποσύρουμε και επίσης ε, συμφωνούμε απόλυτα με τη συμβαστική τροπολογία 12 με την ε, διατύπωση που έχει αποκρισταλωθεί. Έχουμε κάποιες προτάσεις όμως για τροποποίηση της ε, συμβαστικής τροπολογίας 11. Και θα ήθελα να ρωτήσω ε, αν γίνεται να περιλάβουμε στην έκθεση το καθεστώς ουδετερότητας με μερικών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χαίρομαι γιατί στην τελευταία εκδοχή συμπεριλήφθηκε και το θέμα αυτό στη συμβαστική τροπολογία 11. Θα ήθελα και στη συμβαστική τροπολογία πάλι 11 να, να τροποποιήσουμε μία λέξη και που λέει με την ανάπτυξη των στρατιωτικών ικανοτήτων και που λέει ανάπτυξη, θα ήθελα τη λέξη ανάπτυξη, το development να το πούμε deployment. Νομίζω ότι θα συμφωνήσει ο κύριο Έλερ το development να γίνει deployment. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 124 θα ήθελα να ζητήσω ψηφοφορία κατά τμήματα. Να πούμε χαίρετε για την ανοιχτή συζήτηση μέχρι όπως προβλέπει το άρθρο 42.3 και το δεύτερο τμήμα ζητά από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστούν τον ορισμό μιας γνήσιας ε, βιομηχανικής ε, αμυντικής πολιτικής ε, που θα ευθυγραμμίζεται με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτά τα δύο τμήματα θα ήθελα να ψηφίσουμε ξεχωριστά. Κατά του λοιπού είναι αρκετά καλή έκθεση. Όπως σας είπα, ο εισηγητής κατόρθωσε να συμπεριλάβει στην έκθεσή του πολλέ από τι τροπολογίε, όχι μόνο των σοσιαλιστών, αλλά και τροπολογίε σχεδόν όλων των πολιτικών ομάδων. Πρόκειται για μια έκθεση που για πρώτη φορά άπτεται ενό πολύ σοβαρού θέματο και το χειρίζεται με πολύ σοβαρό τρόπο. Και χάρη στην έκθεση αυτή και στην συνεννόηση και συνεργασία που είχαμε. Ελπίζω ότι θα εγκριθεί εμεί πάντω ότι την υπερψηφίσουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Σα ευχαριστώ, κύριο Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση όσον αφορά αυτά τα δύο, ε, το ε, στρατιωτικό προσωπικό και το μη στρατιωτικό. Κοιτάξτε, εγώ έχω την εντύπωση ότι ειδικά το στρατιωτικό προσωπικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη, αδιαμφισβήτητα εφαρμόζει τις επιταγές της πολιτικής. Δηλαδή, ό,τι εντολή τους δώσουν οι πολιτικοί, την δέχονται και την εφαρμόζουν στην πράξη. Ε, όσον αφορά τώρα την εμπειρία με την Κομισιόν, ίσως ε, σε κάποια επίπεδα της ε, Κομισιόν να υπάρχουν εκεί στελέχοι που να διαφορούν παντελώς τι θέλει ο Επίτροπος ή το πολιτικό επίπεδο αυτοί κάνουν ε, αυτό που επιθυμούν εκείνοι διαφορετικό είναι αυτό εγώ έχω την εντύπωση την πολιτική ότι στον μη στρατιωτικό τομέα, στην ε, Κομισιόν, αυτή η αυτονομία είναι πολύ μεγαλύτερη από την ε, πολιτική βούληση, την εκάστοτε πολιτική βούληση. Γι' αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται να ανησυχούμε ότι το στρατιωτικό σκέλος ε, δεν θα εφαρμόσει ε, την πολιτική βούληση. Οι στρατιωτικοί το έχουν συνηθίσει αυτό. Στην διοίκηση εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει μια δικιά της δυναμική. Εκεί πράγματι έχουν εντύπωση ότι τα στελέχη της Κομισιόν δεν κάνουν πάντα αυτό που επιθυμούν οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι. Ε, Κυρία Γιατανμάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να επενέσω τον εισηγητή για την έκθεσή του που είναι πολύ καλή παρόλο που θα προτείνω τροπολογίες. Μόλις έλαβα τις συμβαστικές τροπολογίες δεν πρόλαβα να τις διαβάσω. Θέλω να έχω λίγο χρόνο για να τις εξετάσω πολύ προσεκτικά. Δεν πρόκειται να σχολιάσω τώρα. Έχω κάποια σχόλια. Η έκθεση αυτή δίνει έμφαση, υπερβολικά κατά τη γνώμη μου, στην στρατιωτική πτυχή, στο στρατιωτικό σκέλος. Όταν λοιπόν εγώ διαβάζω την έκθεση Έλερ. βλέπω μια ανισορροπία. Θα ήθελα να γιατί η εντύπωση που αποκομίζω διαβάζοντα την έκθεση είναι ότι ο εισηγητή είναι υπέρ τη στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων και όχι υπέρ τη πολιτικο-στρατιωτική. Θα πρέπει να εξορροπηθεί αυτή η έκθεση, ενισχύοντα λίγο το πολιτικό σκέλο, όπω είναι ενισχυμένο και το στρατιωτικό. Επίση, γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει μία κρίση. Δεν έχει αρκετό προσωπικό δεν μπορεί να στελεχώσει αυτές τις μονάδες. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα κάνει στις αρχές του 2012, γιατί τα κράτη-μέλη δεν έχουν καταθέσει τις εισφορές τους ακόμη. Δεν υπάρχουν πόροι. Και είπαμε ότι είναι σημαντικό να προβάλλεται εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνεται ορατή. Το πιο σημαντικό όμως τώρα είναι να εξασφαλίσουμε αρκετούς πόρους και ικανότητες για να μπορέσουμε να στείλουμε αυτά τα στρατεύματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λόζινγκ. Πρέπει να πω ότι ορισμένες απόψεις με εκπλήσουν η δική μου στάση απέναντι σε αυτή την έκθεση δεν νομίζω θα σε εκπλήξει. Εγώ λοιπόν επιθυμώ να αναφέρω κάποια θέματα που προέκυψαν από τη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή κατακλυζόμεθα από σκάνδαλα που έχουν σχέση με στρατιωτικές ενέργειες. Και ε, ο κύριος Εγκαλά λέει ε, τουλάχιστον εγώ έτσι το κρίνω, αφελή πέστε με, λέει λοιπόν ότι το, στρατιωτική συνδέονται άμεσα με την πολιτική βούληση. Λέξη κλειδί, κούντους. Πού ήταν η πολιτική βούληση? Κατά τη δική μου λοιπόν άποψη και κατά την άποψη πολλών άλλων, μια στρατιωτική επιχείρηση πάντα ενέχει τον κίνδυνο της ε, ανεξαρτητοποίησης και πάντα εγκυμονεί ο κίνδυνος σε τέτοιου είδου ε, επιχειρήσεις ε, φρικαλαιοτήτων και βίων πράξεων. Σε όλη αυτή τη συζήτηση υπάρχει ένα θέμα που θέλω να το αντιστρέψω. Δηλαδή, γίνεται εδώ η συζήτηση ω ΣΑΝ να επρόκειτο για στρατιωτική υποστήριξη πολιτικής πράξης. Και εδώ θέλω να πω το εξή. Εγώ είμαι σε άμεση επαφή με ΜΚΟ, με την Medico International, ε, με τον Ερυθρό Σταυρό, ε, με την Γερμανική Υπηρεσία των Οργανισμών Ανάπτυξη. Όλοι αυτοί λοιπόν λένε εμεί δεν θέλουμε να έχουμε στρατιωτική προστασία. Τουναντίον, ε, τα καταφέρνουμε μόνοι μα. Το έχω ακούσει και το έχω πει και εγώ επανειλημμένα και θέλω να καταστήσω ένα πράγμα σαφές. Όλη αυτή η συζήτηση για, το, ε, για τους στρατιωτικούς ε, που υποτίθεται, αντίστροφα το λέει η Μιλήτρια, η πολιτική που στηρίζουν τους στρατιωτικούς, αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Αυτό που ενδιαφέρει είναι πολιτική υποστήριξη στρατιωτικών επεμβάσεων και επιχειρήσεων. Ας δούμε κατά το παρελθόν τι ακριβώς συνέβη. Είμαι πεπισμένη ότι η επιδιωκόμενη συνεργασία στρατιωτικών και πολιτικών όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ οφείλεται στο ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να χρηματοδοτηθούν, δεν υπάρχουν χρήματα και γι' αυτό θέλουν να συμπεριλάβουν και τους μη στρατιωτικούς. Αλλά Πρόκειται καταρχήν για ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που βασίζονται σε εξισορρόπηση συμφερόντων και άσκηση εξουσίας. Αυτή η συζήτηση δεν γίνεται. Και αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οτιδήποτε αναφέρεται εδώ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κάτω από διαφορετικό πρίσμα. Ας πάμε τώρα στην έκθεση. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα σημείο στην έκθεση αυτή όπου να μην θέλουμε να καταθέσουμε ουσιαστικές τροπολογίες. Ήδη κατά την ανταλλαγή απόψεων κατά τέλη Σεπτεμβρίου είπα τη γνώμη μου και δεν χρειάζεται να την επαναλαμβάνω λεπτομερώς. Οι τροπολογίες που έχουν κατευθεί χρήζουν βελτιώσεων ε, έχουν γίνει κάποιε βελτιώσει, κατά την άποψή μα όμως όχι επαρκή. Και όσον αφορά την κατεύθυνση που επιθυμώ εγώ και η πολιτική μου ομάδα, δεν ακολουθούν οι τροπολογίε στην κατεύθυνση αυτή. Ως εκ τούτου εγώ και η πολιτική μου ομάδα, επουδενή δεν θα συμφωνήσουμε με τις τροπολογίες αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριο Γουαλτιέρη. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σύντομα. Ήθελα μόνο την εκτίμησή μου να εκφράσω για την ε, δουλειά του εισηγητή. Ε, όλη την προσπάθεια που κατέβαλε για τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες, νομίζω με μεγάλο πνεύμα συνεργασίας, τη συνέταξε και πραγματικά νομίζω ότι μπορεί να συμφωνήσει κανείς. Δεν θέλω να υπησέλθω. ήδη τα είπε όλα ο εισηγητής και κάποιοι από τους παρεμβαίνοντες. Ιδιαίτερα για το ζήτημα της ισορροπίας μεταξύ του στρατιωτικού και του πολιτικού και της εξωτερικής παρέμβασης. Τώρα, όσο αφορά την τροπολογία 24, 124, Ίσως το πρόβλημα είναι να διευκρινίσουμε περισσότερο το δεύτερο τμήμα, γιατί θα μπορούσε να δώσει την εντύπωση ότι αναφέρεται στην έρευνα για την, στην έρευνα για την άμυνα και ίσως αυτό θα ήταν μια πολύ έντονη διατύπωση και καταλαβαίνω πώς το βλέπει ο εισηγητής. Θα μπορούσαμε ίσως να διευκρινίσουμε ότι παραπέμπει στην σε μια πολιτική της αγοράς, της Ευρωπαϊκής Άμυνας για την συνένωση αυτών των υποδομών, δηλαδή για την αμυντική βιομηχανία. Ίσως λοιπόν η διατύπωση της τροπολογίας μοιάζει να συνδέεται περισσότερο με το ζήτημα της στρατιωτικής έρευνας ε, για το πρόγραμμα πλαίσιο, ε, το, περισσότερο σαν να παραπέμπει στη δυτή φύση παρά στη στρατιωτική φύση. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ του προγράμματος ε, του προγράμματος πλαισίου, όπως λέει και η συμβαστική πρόταση 10, και να διαχωριστεί το άλλο ζήτημα που αφορά τη συνεργασία πολιτικού στρατιωτικού. Θέλουμε να προάγουμε την ανάπτυξη μιας ε, διαδικασίας ανάπτυξης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Πρέπει να ξεκαθαριστούν αυτά τα δύο. Ευχαριστώ. Ε, εγώ θα να εγκομιάσω την ε, θαυμάσια έκθεση του εισηγητού και να τον ε, επενέσω για το διαλλακτικό του πνεύμα και την προθυμία του να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερες τροπολογίες στις ε, πολύ καλές του συμβιβαστικέ προτάσεις. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική στη φάση που βρισκόμαστε. Δεν θα πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να δώσουμε μια όθηση σε ζητήματα που μπορεί να είναι επίμαχα, αλλά που ακριβώς εξαιτία της χρηματοπιστωτικής χρήσης, αυτές οι, συνεργα... αυτές οι συνεργασίες είτε οι πολιτικοστρατιωτικές, είτε σε επίπεδο επένδυση στην έρευνα, είναι σημαντικές. Πιστεύω επίσης και φυσικά διαφωνώ με εκείνους που έχουν μια αρνητική προκατάληψη για το ρόλο των στρατιωτικών. Άλλωστε και στη δική μου έκθεση που πριν από λίγο συζητήσαμε διαπιστώνω την κεφαλαιότητη σημασία που έχει ο στρατιωτικός κλάδος, ο στρατός για την βοήθεια του άμαχου πληθυσμού, είτε σε περίπτωση ε, ε, ανθρωπιστικής καταστροφής, είτε για άλλους, άλλες καταστροφές όπως είναι οι επιθέσεις με υλικά, χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά, πυρηνικά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαρθρώσουμε καλύτερα τη συνεργασία μεταξύ των πολιτικών και των στρατιωτικών ικανότητων γιατί ο στρατός είναι που έχει πολύ μεγαλύτερες ικανότητες σχεδιασμού και προγραμματισμού και πολύ πιο πλούσιες γνώσεις για ουσίες χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές, για παράδειγμα, κάτι που ο πολιτικός κλάδος δεν διαθέτει. Ή είναι πολύ αποσπασματικές οι πληροφορίες, η γνώση που έχει. αποσπασματικέ και είναι πληροφορίε οι γνωσει που εχει συνεργασία. Και ειναι σημαντικη κερια η πολιτικο-στρατιωτική είναι και το ευρωπαϊκό ατού. Είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διαπιστώσαμε ότι στις μεγαλύτερες καταστροφές χρειάστηκε να αναπτύξουμε και στρατιωτικές δυνάμεις. Αν μη τι άλλο, για να εξασφαλίσουμε την άφηξη της ε, βοήθειας στους δικαιούχους, στον πληθυσμό που, τη χρειαζόταν. Πριν από λίγο, η κυρία Πράντνερ μίλησε γι' αυτό. Ε, ε, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα πεδία μάχης, κάτι που δεν γίνεται. Και να τα χρησιμοποιήσουμε τα πεδία μάχης και για τις ε, προσπάθειες ενέργειας ανακούφισης ε, της κρίσης, για την επισητιστική βοήθεια, ε, ανθρωπιστική συγγνώμη, βοήθεια και το καθεξής. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και το δόγμα μας αυτό της στρατιωτικής επέμβασης θα πρέπει να προστατεύσουμε τους ε, πολιτικούς πληθυσμούς είτε σε περίπτωση ανθρωπιστικής καταστροφής είτε σε περίπτωση περιβαλλοντικής, οικολογικής καταστροφής είτε στην περίπτωση καταστροφής ε, όπως αυτές, αυτές που βρίσκουμε στο Κονγκό, τις γυναίκες που είναι θύματα βίας. Φυσικά οι ομάδε κρούς ήταν πριν από λίγο που έλεγε Battlefield στη συγγήτρια και όχι τα πεδία μάχη. Πιστεύω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα. Το βλέπουμε αυτό σε όλου του τομεί και πριν από λίγο το είδαμε ξεκάθαρα και στον τομέα του διαστήματο, τη πολιτική διαστήματο. Αυτά και συγχαρητήρια, η έκθεση είναι καταπληκτική. Ευχαριστώ, κύριος Έλλερ. Ähm, ähm, Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω το εξής. Αφενός αναφέρθηκε ότι ε, θα πρέπει να υπάρχουν αριθμοί, δηλαδή ε, πόσες είναι οι στρατιωτικές και πόσες οι μη στρατιωτικές επεμβάσεις. Κοιτάξτε, εγώ κατέθεσα ένα έγγραφο όπου υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Νομίζω, νομίζω όμως ότι ήταν λάθος τώρα την έκθεση να την βασίσουμε μόνο σε στοιχεία γιατί θα πρέπει να εκφράζει την άψη του Κοινοβουλίου και μετά από ένα και δύο χρόνια. Και τι γίνεται μετά από ένα-δύο χρόνια μπορεί να έχουν προσθεθεί και μια-δυο περισσότερες ε, πολιτικές επιχειρήσεις, άλλες στρατιωτικές. Αν λοιπόν τώρα βασιστούμε μόνο σε μεμονωμένους αριθμούς για να στηρίξουμε ένα πολιτικό σκοπό, αυτό είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο για την έκθεση, κυρίως κάτω από το πρίσμα ότι η έκθεση δεν θα είναι επίκαιρη. Όσον αφορά τα battle groups, τις ομάδες κρούσης, θεωρώ ότι υπάρχουν πράγματι στρατιωτικές δυνατότητες των κρατών μελών Υπάρχουν και δυνατότητες πολιτικής προστασίας στις καταστροφές και η έκθεση λέει ότι και τα δύο αυτά όργανα ή εργαλεία είναι ισότιμα και δεν αμφισβητείται αυτό. Σε ορισμένα σημεία προσπαθούμε να πούμε ποιες είναι οι ανάγκες μας, για ποιες αποστολές και για ποιους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι δεν ισχύει αυτό που ελέγχθη ότι ε, δεν ασχολούμεθα θεπαρκώς με το μη στρατιωτικό κομμάτι. Όχι, εμείς καλούμε ξεκάθαρα τα κράτη-μέλη να ε, διαθέτουν περισσότερο προσωπικό για πολιτικές καταστροφές, είτε και στρατιωτικούς είτε και μη στρατιωτικούς. Ε, λέμε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να εγκρίνουμε τον ένα στόχο μετά τον άλλο και μετά στην πραγματικότητα, στην υλοποίηση των στόχων να μην έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια. Γιατί στην περίπτωση αυτή Κατ' ουσίαν τι κάνουμε. Ε, επισημαίνουμε στα κράτη-μέλη ανάμεσα στις αποφάσεις και την εφαρμογή τους. Οι battle groups, κατά την άποψή μου, δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ για πολιτικούς σκοπούς. Αλλά τι γίνεται ανάμεσα μάλλον στο φάσμα των δυνατοτήτων που υπάρχουν, ε, μία ομάδα κρούση, ένα battle group, πρέπει σε μία στρατιωτική επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα αργότερα να συνεργαστεί περισσότερο με πολιτικές αποστολές. Αυτό είναι το όλο θέμα. Όχι ότι οι battle groups από μόνες τους ε, θα εντάσσονται μέσα σε πολιτικές επιχειρήσεις. Και καθαρά λειτουργικά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Απλά να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες και οι ε, battle groups όπως σας είπα να συμμετέχουν. Όσον αφορά το ερώτημα στρατιωτικό ή ε, πολιτικό προσωπικό. Νομίζω ότι στις επαφές που είχα με τις διάφορες δομές ε, ποτέ δεν βίωσα αμοιβαία δυσπιστία. Κάθε άλλο όλοι ενδιαφερόντουσαν για το στόχο της επιχείρησης και τις επιχειρησιακές ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ ε, που όπως και σε άλλους τομείς δεν βασιζόμαστε μόνο στην αναλογία και στην ισορροπία αλλά λέμε με απόλυτα σαφήνεια ε, και αυτό αφορά αυτό που είπε και ο συνάδελφος Ντοζόν και άλλοι, ότι όσον αφορά αυτή την σχέση του στρατιωτικού και μη στρατιωτικού προσωπικού, εμείς λέμε στα αγγλικά επισημαίνει την ανάγκη αμοιβαίου σεβασμού ε, του στρατιωτικού και μη στρατιωτικού ρόλου όπως επίσης και τους στόχους για να καταστήσει σαφές ότι ε, θα υπάρχει ένας σωστός συγκερασμός δυνάμεων που θα διατίθεται κατά περίπτωση. Και αυτό είναι τέλος της παράθεσης. Νομίζω λοιπόν ότι αντί να κάνουμε εδώ ιδιαίτερα ιδεολογικά φορτισμένες συζητήσεις να ασχολούμαστε με την πράξη να αποφύγουμε ε, το να υπάρχει αριθμητική εξισορρόπηση. Εμείς έχουμε στόχους. Αυτό που καλούμεθα να κάνουμε είναι να εκπληρώσουμε τους στόχους και όχι να λύσουμε μαθηματικές εξισώσεις. Άρα δηλαδή ίδια σημασία τόσο για το στρατιωτικό όσο και για το μη στρατιωτικό σκέλος. Και ένα τελευταίο θέμα, επειδή θίγεται επανειλημμένα και πρέπει να σας πω και καθαρά πολιτικά ότι είναι απαράδεκτο. Κοιτάξτε, εσείς αναφέρεστε στις ΜΚΟ, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ας πούμε στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Δεν είναι αλήθεια αυτό που είπατε. Εμείς συζητήσαμε με πολλές από αυτές τις ΜΚΟ και βεβαίως οι οργανισμοί αυτοί λένε ότι για την δική μας την επιχείρηση δεν χρειαζόμαστε ε, στρατιωτική υποστήριξη. Αλλά λένε όμως, εντάξει το λένε αυτό, αλλά λένε και από την άλλη ότι εμείς δεν μπορούμε καν να αναπτύξουμε τις δραστηριότητες μας σε μια περιοχή αν δεν νιώθει ασφάλεια ο πληθυσμός, οι πολίτες. Ε, δεν μπορεί να επέμβει ένας γιατρός όταν κινδυνεύει η ζωή των ανθρώπων, όταν υπάρχει κίνδυνος γενοκτονίας. Κανένας λοιπόν από αυτούς τους οργανισμούς δεν αμφισβήτησε ότι στον Ταφούρ ή και σε άλλες περιοχές καταρχήν είναι απαραίτητο από στρατιωτική σκοπά, σκοπιά να ε, διασφαλιστεί η ασφάλεια να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι γιατροί. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ε, απορρίπτω κατηγορηματικά αυτό που λέει η κυρία Λόιζινγκ ότι η ΜΚΟ, ε, μάλλον τι κάνει κύριε Λέζινγκ, παίρνει ως όμοιρους ε, στην επιχειρημα, επιχειρηματολογία της, ε, της ΜΚΟ, της χρησιμοποιεί της ΜΚΟ, εμείς δεν συμφωνούμε γιατί σας είπα μιλήσαμε με αυτές τις ΜΚΟ. Τελειώνοντας λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, νομίζω ότι από κοινού καταβάλαμε την προσπάθεια να δώσουμε ηχηρή φωνή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τη, βάση όπου, από τη φάση που βρισκόμαστε τη σύνταξη ε, των ε, συμβαστικών προτάσεων. Ε, Βεβαίω και γνωρίζω ότι υπάρχουν αντιδράσει και από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλου όσοι συνέβαλαν επικοδομητικά στη σύνταξη τη έκθεση αυτή. Και θέλω να σα πω ότι η ιδεολογική επιχειρηματολογία δεν θα βοηθήσει του ανθρώπου, δεν μπορεί να του βοηθήσει προσφέροντα ιδεολογία. Συγκεκριμένα πράγματα χρειάζονται επιτόπου οι άνθρωποι αυτοί. Σας ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε την Πέμπτη το πρωί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη γνωμάδα της κυρίας Λέζινγκ για τα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά τις επιθέσει μάλλον από τέτοια όπλα και την έκθεση Έλερ. Άλλα θέματα υπάρχουν για τα διάφορα. Όχι, οπότε ραντεβού αύριο ε, στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και την Πέμπτη για την ψηφοφορία. Η επόμενη μας ε, συνεδρία θα γίνει στι 15 Νοεμβρίου, 3 το απόγευμα, με δύο προσκεκλημένους, τον ε, στρατηγό Βαμπό, που είναι νέο γενικό διευθυντή του Στρατηγικού Αρχηγείου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να θέσουμε και αυτό το ζήτημα στο στρατηγό, ε, στα πλαίσια των δράσεων τη ΕΠΑ. Και ο κύριο Σιμόνοβιτ, που είναι ο Κροάτη Υφυπουργό Άμυνα, επιφορτισμένος με διεθνή και ευρωπαϊκά ζητήματα. Αυτή η δύο ψηλή προσκεκλημένη μας στην επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.